Good uh, Συνάδελφοι, καλησπέρα, τουλάχιστον όσοι είναι παρόντες. Θα ήθελα να εγκρίνω το σχέδιο ημερησίας διάταξης σε πρώτη φάση και αν δεν έχετε αντιρρήσεις, ε, θεωρείται εγκεκριμένη η ημερησία διάταξη. Πολύ ωραία. Να εγκρίνουμε επίσης τα πρακτικά της ε, συνεδρίασης, των συνεδριάσεων μάλλον, μεταξύ 25 Σεπτεμβρίου και 19 Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, αντιρρήσει, παρατηρήσει, τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα. Και σα ευχαριστώ. Καμία ανακοίνωση σήμερα από πλευρά του Προέδρου. Στο σημείο 4 όμω θα σα πω πώ πάνε οι διοργανικέ διαπραγματεύσει. Τρει στον αριθμό σε τρεις περιπτώσεις έχουμε λευκό καπνό. Για να κάνω και μία αναφορά στο Βατικανό και στον Πάπα. Άρα, λοιπόν, τρεις τριμερείς διαλόγους, ε, τριμερείς ε, διαλόγους ολοκληρώσαμε τελικός ε, διάλογος για τις μεταβατικές ρυθμίσει που έλαβε χώρα στις 25 Οκτωβρίου Και όπω ξέρετε ήταν διαδικασία fast track ταχεία διεκπαιρέωση για το CRD package και στον τρεμερή διάλογο καταφέραμε να φτάσουμε σε πολιτική συμφωνία με βάση συμβιβασμού ότι οι χρήστες θα χρησιμοποιηθεί μάλλον καταρχάς το κείμενο του Συμβουλίου και θα αφαιρέσουμε τα δυναμικά στοιχεία από 20% σε 0%. Για τη μεταβατική φάση δεν υπήρξαν σημαντικές ε, διαφορές. Διαβουλεύσει για την Επιτροπή προβλέπονται για 20 και 21 Νοεμβρίου. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί οι διατάξει θα τεθούν σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου και ω εκ τούτου θα έχουμε επαρκή χρόνο μέχρι την νόμιμη θέση σε εφαρμογή της σταδιακής αυτής ε, υλοποίησης προκειμένου να είναι σταδιακή αυτή η προσαρμογή στα πιο αυστηρά λογιστικά πρότυπα. Δεύτερο τρίμερη διάλογο σε ό,τι αφορά την σχετική ιεράρχηση ήταν πολύ κοντινέ και οι θέσει του Κοινοβουλίου. 25 Οκτωβρίου λοιπόν καταφέραμε να φτάσουμε σε συμφωνία, στην πρώτο τριμερή διάλογο και στις 21 Οκτωβρίου διανεμήθηκαν οι τελικές ε, θέσεις και ε, έτσι δημοσιεύθηκε η πρόταση για την υλοποίηση σε μεταφορά σε εθνικό δίκαιο σε ό,τι αφορά και τα θέματα των παραγόγων σε ό,τι αφορά θέματα των προτιμήσεων ε, σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη τους σε λογική σκέψη η συμφωνία λοιπόν επιτεύχθηκε μετά από πολλοί σε διαλόγους για το σχεδιο ΕΦΣΑ FC2. Δύο θέματα παραμένουν εκκρεμή σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση δεν ολοκληρώθηκε αυτό μετά τον τελευταίο τριμερή διάλογο, γιατί θα το ανοίξει εκ νέου το θέμα αυτό το Συμβούλιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πετύχαμε καλό συμβιβασμό. Και η θέση συνάδει με τα όσα είχαν συμφωνηθεί από πλευρά του Κοινοβουλίου. Και φυσικά αυτό το αποτέλεσμα, πολύ ικανοποιητικό, αποτελεί μια καλή είδηση προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το 2018. Από αρχές 2018 υπάρχει και μια νομική βεβαιότητα για τους ε, επενδυτές. σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των επενδύσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα θέματα αυτά λοιπόν του τριμερίου διαλόγου ήταν πάρα πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά το, τα δάνεια. Αυτοί οι τριμερείς διάλογοι λοιπόν εστέφτησαν με επιτυχία. Ήταν μια στιγμή καλή για το Κοινοβούλιο. Έγκυρα και τα αποτελέσματα για να προσαρμοστεί. Και ας περάσουμε λοιπόν στο σημείο 5 της μερικής Έγκριση του σχεδίου χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων της Επιτροπής Οίκων για το 2018. Θα βρείτε στους φακέλους σας τα... τις ημερομηνίες που πρότειναν και ενέκριναν οι συντονιστές της 26 Οκτωβρίου αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το πέρας της σημερινής συνεδρίασης, το σχέδιο αυτό θα θεωρηθεί εγκεκριμένο. Το σχέδιο χρονοδιαγράμματος. Πολύ ωραία. Και να περάσουμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διατάξης ε, της έκθεσης σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η συγητή μα είναι αυτή τη φορά. Ξέρετε ότι πρόκειται για γνωμοδότηση άλλωστε, γιατί ε, το έχουμε εκπεριτροπής με την ε, Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Είναι λοιπόν η σειρά μας να γνωμοτήσουμε στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Λούτε Κρίνερ Μάιερ, ο εισηγητής μας. Είμαστε στη φάση εξετασής των τροπολογιών. 104 τροπολογίες λάβαμε. Και ο εισηγητής λοιπόν έχει το λόγο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για συζήτηση, αλλά νομίζω ότι θα επαρκέσει. Όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, πρόκειται για μια γνωμοδότηση σε μια έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ο εισηγητής της γνωμοδότησης είμαι εγώ. Και ξέρετε ότι θεωρώ ότι δεν πρέπει η γνωμοδότησή μας ε, να έχει παραπάνω από 1500 λέξεις. Με καλές τροπολογίες μπορούμε να εμπλουτίσουμε το αρχικό μας κείμενο. Είπατε ότι έχουμε πάνω από 100 τροπολογίες. Από αυτές τις τροπολογίες προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τις πιο σημαντικές που οδηγούν προς την ίδια κατεύθυνση, που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ε, προτείνουμε 16 συμβαστικές τροπολογίες που θα εξεταστούν για πρώτη φορά αύριο στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Επιπλέον προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και υποστήριξη για κάποιες βασικές τροπολογίες. Θα σας αναφέρω κάποιες βασικές τροπολογίες. Καταρχάς, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι να δρά στους τομείς που αποτυγχάνουν οι αγορές και να υποστηρίξει τους βασικούς τομείς προτεραιότητας το, της α, οικονομικής πολιτικής, παραδείγματος τη χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας, ε, την υποστήριξη της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, υποστήριξη σε, σε χρηματοδότηση, κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερο σημείο που θέλουμε να τονίσουμε στην έκθεση είναι η ανάγκη να τονίσουμε, την, να δούμε τι, πώς θα επηρεάσει το Brexit τη χρηματοδοτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Τραπέζας Επενδύσεων. Επίσης, τις τελευταίες ε, μέρες είδαμε ότι υπάρχουν σημαντικά οικονομικά θέματα, παραδείγματος χάρη ε, πρόληψη φορολογικών απατών, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, ε, ξεπλήματος χρήματος που μπορούν να συνδεθούν με κάποιες δραστηριότητε πελατών της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων. Επίση, θα τονίσουμε τη σημασία να υπάρξει μία εντολή για την εξωτερική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δηλαδή τη χρηματοδότηση στο εξωτερικό, και να χρηματοδοτήσουμε βασικέ οικονομίε του εξωτερικού, όπω η Ουκρανία, παραδείγματο χάρη. Περιμένω λοιπόν τη συνάντηση των σκιωδών αύριο και ελπίζω να υπάρξει συνένεση για τι τροπολογίε και για τι μεμονωμένε τροπολογίε που έχουν κατατεθεί. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή. Περνάμε στους κοιόδες εισηγητές. Ο κύριος Ραμόν Χαουρέγγι Ατόντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, ευχαριστώ τον κύριο Νίντερ Μάγερ για τη δουλειά που έκανε. Απλώς μια ματιά έριξα στο κείμενο. Ε, που μας έφερε για τη συνεδρίαση το πρωί του Σαββάτου και βλέπω ότι υπάρχει βούληση να λάβει υπόψη του πολλές από τις τροπολογίες που κατέθηκαν. Εγώ θα περιοριστώ στο να εξηγήσω τι παρουσίασε η σοσιαλιστική ομάδα. Καταρχάς, υπάρχει μεγάλη σημασία στη μακροοικονομική ε, μεγάλη σημασία που δίνεται μάλλον για την ε, μακροοικονομική επίπτωση της δουλειάς που κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι προβλέψεις για μακροοικονομικές επιπτώσεις της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μέχρι το 2020 είναι ε, γύρω στο 2,25% του ΑΕΠ της Ένωσης και μπορεί να δημιουργήσει πάνω από 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε τη μακροοικονομική επίδραση, επίπτωση αν θέλετε, της τράπεζας. Επίσης, μια διαφορετική απόχρωση από αυτή του εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποτίθεται ότι εξακολουθεί να έχει μια αντικυκλική δραστηριότητα. Ε, δηλαδή, ο όγκος των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει φτάσει στο επίπεδο των επενδύσεων που είχαμε πριν από την κρίση. Ακόμα. Και επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που η τράπεζα έχει καθώς τονώνει την ανάπτυξη και τη ζήτηση, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε. Επίσης, υπάρχει μια τροπολογία από τους σοσιαλιστές για την ανάγκη να διευκρινίσουμε κάποιες αναφορές στον αριθμό των εντολών που θεωρεί ο εισηγητής ότι είναι υπερβολές, δηλαδή πολλές υπερβολ... διαφορετικές χρηματοδοτήσεις. Καλύτερα να μην μιλήσουμε για εντολές, mandates. Γι' αυτό προτείναμε να διαγράψουμε αυτή την παράγραφο που κάνει λόγο γι' αυτό. Επίσης, θεωρούμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για τη σημασία της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε εξωτερικό επίπεδο, εξωτερικέ δραστηριότητες. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση για την συνεργασία και αυτή είναι μια αναπτυξιακή τράπεζα. Επίσης πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα πρέπει να κάνει μια αναλυτική δουλειά και να μην λειτουργεί μόνο σαν χρηματοδότης ας πούμε, αλλά και σαν τράπεζα γνώσεων ε, όπου συλλέγονται καλές πρακτικές ε, και χάρη στους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, να τονίσουμε τη σημασία του να ενισχύσει τις δραστηριότητες η τράπεζα στο επίπεδο της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τις δεχτεί αυτές τις τροπολογίες ο εισηγητής. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητα παίζουμε την το τεχνολογικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι άλλε χώρε όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε μας ξεπερνάνε κατά πολύ. Επίση, κάποιε άλλε τροπολογίε που έχουμε υποβάλει και έχουν σημασία για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μια ειδική αναφορά στην δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για έργα τα οποία έχουν δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Επίσης, το Brexit να μην οδηγήσει σε μείωση του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σημαντικό αυτό, στον αγώνα που κάνει η τράπεζα κατά της φοροδιαφυγής. Υπάρχουν πληροφορίες ε, για φορολογικές ε, απάτες που προκαλούν που έχουν φοβερό αντίκτυπο ας και κινητοποιούν ε, την ε, κοινή γνώμη, δημιουργούν μάλιστα πολλέ ανησυχίε, α πούμε τα Panama Papers. Ε, παίζει ρόλο εκεί η τράπεζα. Επίση, στον τομέα του πολιτισμού έχει μεγάλη σημασία ο ρόλο τη τράπεζα με τι επενδύσει που κάνει. Επίση, τη δυνατότητα η τράπεζα να χρησιμοποιήσει τα ομόλογα σε στενότερη σχέση με τους πολίτες Δηλαδή να, να βγάλει, να εκδώσει ας πούμε ομόλογα ας πούμε και έτσι να αυξήσει την, τα κεφάλαια ας πούμε. Τέλος, υπάρχει μια τροπολογία που ενδιαφέρει τους σοσιαλιστές, τη δυνατότητα δηλαδή τα ωφέλη τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τα κέρδη, τα έσοδα, ας πούμε, να συνυπολογίζονται στον κοινοτικό υπολογισμό και σε ό,τι αφορά τι επενδύσει των κρατών, οι συνεισφορές των κρατών μελών σε δημόσια έργα να μην ε, συνυπολογίζονται στο έλλειμμα, στα ελλείμματα, στα ελλείμματά τους. Έτσι. Αυτές οι τροπολογίες των σοσιαλιστών θα δουλέψουμε με τον εισηγητή, ούτω ώστε να φτιάξουμε την πιο συνενετική, όσο να τον περισσότερο συνενετική δηλαδή γίνεται, ε, γνωμοδότηση γίνεται. Ευχαριστώ. Ποιο είναι ο σκιώδη ηγητή του ΙΣΙΑ, δεν νομίζω ότι είναι εδώ. Από του ε, φιλελεύθερου, ούτε. Έχουμε, ούτε εδώ έχουμε σκιώδη. Η κυρία Σκοτ Κέιτ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι πολύ που οι σκιώδε εισηγητές δεν βρίσκονται εδώ. Ελπίζουμε να υπάρξουν αλλαγές. Θα δούμε και τις τροπολογίες σήμερα λίγο αργότερα και το τι προσπαθούμε να επιτύχουμε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι χαίρομαι πολύ που πολλές τροπολογίες που προτείναμε εγκρίθηκαν και οι συμβιβασμοί προσθέτουν θετικά αποτελέσματα στο κείμενο. Χαίρομαι που οι συνάδελφοι συμφωνούν ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε σε αυτήν την Επιτροπή την ευκαιρία να επιμείνουμε στην σημασία της ενίσχυσης των επενδύσεων προκειμένου να επωφεληθούν οι ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της έλλειψης επενδύσεων των τελευταίων ετών. Και θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή το ΕΦΣΥ δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι παραμένουν αναπαρκείς οι επενδύσεις ε, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Είναι σημαντικό να αναλάβουμε δράση προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να υποστηριχτεί η, ανάπτυξη, η βιώσιμη ανάπτυξη. Διαφωνούμε στο κείμενο με το γεγονός ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί ε, προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία πως ε, η δημοσιονομική εξυγίανση έχει πλήξει την ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να βρεθεί συμφωνία σε αυτό το τομέα. Είναι μια μόνιμη δυσκολία που έχουμε ανάμεσα στις ομάδες μας. Θα ήθελα ο εισηγητής και οι σκιώδες εισηγητές να δώσουν σημασία στα εξή. Το στόχο του 1,5% και της επένδυσης στα ορυκτά καύσιμα είναι πολύ σημαντικό μιας και η ε, οι επιστήμονες λένε τώρα ότι προβλέπεται αύξηση θερμοκρασίας κατά 3, βαθμού. βαθμούς. Πρέπει να δεσμευτούμε λοιπόν σε μία αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του Brexit, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει να τηρεί τις δεσμεύσεις του μέχρι να πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στη συνέχεια θα πρέπει να τηρήσει τις, απαιτήσει ε, ε, ε, όποιες απαιτήσεις θα έχουν συμφωνηθεί. Επίσης, θα θέλαμε οι σκιώδεις εισηγητές να δώσουν σημασία στις τροπολογίες 103 και 104 και θα θέλαμε να συμπεριληφθούν αυτές στις συμβιβαστικές προτίσεις. Σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δρά προς όφελος όλων των πολιτών. Και αυτό σε μια περίοδο που οι πράξεις ε, των ανδρών βρίσκονται στο επίκεντρο της ε, προσοχής. Χαίρομαι που αυτός ο φάκελος έχει σημειώσει πρόοδο. Ε, λυπάμαι που δεν μπορούμε να συμμετέχουμε αύριο στη συνεδρία. Ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες μας και εύχομαι στον εισηγητή και στους σκιώδες εισηγητής να επιτύχουν το ε, καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο στα πλαίσια της διαδικασίας CatchDI και ως εκ τούτου θα δώσω το λόγο α, στον εισηγητή. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και τους κοιοδησυγητές για τα σχόλια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε καλούς συμβιβασμούς και να δούμε και το πώς ε, θα μπορούσαν όλοι να υποστηρίξουν τις ε, τροπολογίες, κάποιες συγκεκριμένες τροπολογίες, προκειμένου τελικά να υπάρξει σωστή υποστήριξη στο θέμα αυτό από την Επιτροπή Οίκων. Ευχαριστώ πολύ. Το χρονοδιάγραμμα είναι ως εξή. Στις 20 Νοεμβρίου θα ψηφιστεί στην Επιτροπή το θέμα αυτό. Τέλειο από πλευράς χρονική διαμόρφωση και τώρα να περάσουμε στο σημείο 7 στην κοινή συζήτηση για δύο προτάσεις. CCTB κοινή βάση φορολογίας εταιρεών και CCTB, κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρεών. Ω πακέτο φυσικά τα εξετάζουμε αυτά από κοινού. Εξετάζουμε τις τροπολογίες. Τέσσερις, 414 είναι οι τροπολογίες για το, την κοινή βάση φορολογίας εταιριών και 59 του ΣΥΓΙΤΟΥ για την έκθεση στην κυρίου Τάν και 301 για την έκθεση του κυρίου Λαμασούρ. 30 του ιδίου. Όπως ξέρετε, είναι πολύ σημαντική η νομοθεσία αυτή. Θέλουμε να ληφθεί φυσικά σοβαρά υπόψη ε, η γνωμοδότηση αυτή από το Συμβούλιο γιατί ενδεχομένω να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ψηφιακής φορολόγησης. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τους δύο εισηγητές για όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει. Ο κύριος Τάνγκ, λοιπόν είναι ο πρώτος. Επτά λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες και για τη συνεισφορά του καθενός. Ήταν πραγματικά πολύ συναρπαστικές σε ό,τι αφορά τη συζήτηση τώρα αυτή για τις τροπολογίες. Είναι σε καλό χρονικό σημείο αυτή η συζήτηση, γιατί Χτες τα έγγραφα Paradise ε, κατέδειξαν ότι οι ισχυροί και οι πλούσιοι και ο ήρωας της ε, νεότητάς μου, ο Μπόνο, έχει διαφορετικό, έχουν διαφορετικό τρόπο να πληρώνουν τους φόρους τους. Και υπήρχε και πρόταση των Ρεπουμπλικανών να μεταρρυθμιστεί το Αμερικανικό σύστημα φορολόγησης ε, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του εταιρικού φόρου που 35 σε 20%. Το θέμα είναι πώς αντιδράσει η Ευρώπη τώρα μία αντίδραση την οποία συζητάμε εδώ σήμερα είναι ο ευρωπαϊκός ε, φόρος για τις εταιρείε. Θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή αντίδραση γιατί αναφέρεται και στον, στην αρχή της ενιαίας φορολόγησης γιατί στη βάση φορολόγησης αυτής ε, οι εταιρείε θα μπορούν να αποφασίσουν που θα καταγράφουν τα κέρδη τους σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή με την κοινή βάση φορολογίας των εταιριών. Οι χώρες θα είναι αυτές ε, οι οποίες θα καθορίζουν τι θα φορολογείται πού. Και αυτό θα βάλει ένα τέλος ε, στην φοροδιαφυγή. Στην τροπολογία 94, κ. Μακάρθη, τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Κοιτάξτε όμως, εγώ πιστεύω πραγματικά ότι αν εγκριθούν αν εγκριθεί η κοινή βάση φορολογία εταιριών με χώρες όπως η Ελβετία, όπως η Αμερική, θα καταστεί ο κανόνας αυτό και θα καθορίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο το πώς θα γίνει τη φορολόγηση των εταιριών. Και αυτό με τη σειρά του θα αλλάξει και τη φύση του φορολογικού ανταγωνισμού. Όπως σας είπα, θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο σωστό ανταγωνισμό για τις πραγματικές επενδύσει. Και αυτό που είδα από τι τροπολογίε: υπάρχουν διάφορε ομάδε που πιστεύουν και έχουν διαφορετικές απόψεις σε ό,τι αφορά τον φορολογικό ανταγωνισμό. Εμένα η δική μου ομάδα και πολιτική, το πολιτικό μου κόμμα θέλουν μια ελάχιστη, ένα ελάχιστο συντελεστή φορολόγηση με περιθώριο φυσικά να καθορίζεται αυτό από το κάθε κράτος ξεχωριστά. Αυτό που μου λείπει όμως είναι η πρόταση να υπάρχει και ένα δεσμευτικό ε, συντελεστή, ένα ελάχιστο και ένα δωτόριο. Αυτό θα μπορούσαμε να εξετάσουμε. Αυτό που είδα στις τροπολογίες είναι κάποιες προσθήκες σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες, ε, σε ό,τι αφορά την Google, την, ε, το Facebook κτλ έχω κάνει αναλύσεις και έχω συμπεριλάβει και αναλύσεις και έρευνες του ΑΣΑ κτλ. Και ο κ. Ότμας Κάρας έκανε κάποια σχετική αναφορά στην τροπολογία υπερθυμών 47 και 142. Ο κ. Φέρμπερ, ο Μάρκος, λέει ότι η νομοθεσία για τη φορολόγηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και άλλα στοιχεία. Η προσθήκη αυτή θεωρώ ότι θα πρέπει να προωθηθεί από το Κοινοβούλιο. Κατά δεύτερο, δεύτερη προσθήκη. Βιωσιμότητα. Σε ό,τι αφορά την αρχή της Ιουνίου σε Άλλες τροπολογίες τώρα του κ. Μπούλμαν, Μπαρές αλλά και α, άλλων συναντέλφων, ε, ε, θέτουν το θέμα της ε, μείωσης, προσμείωσης ε, βιωσιμότητος, συντελεστή βιωσιμότητος. Αυτό θα πρέπει να λεφθεί υπόψη, θεωρώ. Και ένα στοιχείο το οποίο επίσης θα ήθελα να τονίσω για να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό σύστημα φορολόγηση, χρειάζεται συνεργασία των φορολογικών υπηρεσιών των διάφορων κρατών. Με υποχρεωτική ε, ε, ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τα φορολογικά. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί προπόθεση. τέλο. τροπολογίες για την αρχική πρόταση. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει υποστήριξη μείωση του κατατατού ορίου γιατί να με συμπεριληφθούν δηλαδή και εταιρείε ε, με χαμηλότερο κύκλο εργασιών από 750 εκατομμύρια. Αν χαμηλώσει αυτό το κατόφλι σε πέντε χρόνια μετά από μια θετική αξιολόγηση προτείνεται να μειωθεί σε βάθος δεκαετίας. Είναι σαφής η κατεύθυνση, αν και υπάρχουν διάφορες προτάσεις σε ό,τι αφορά την προθεσμία. Θεωρώ τώρα Ό,τι αφορά την απομείωση των τόκων. Να πω ότι αυτό είναι και εύκολο να εφαρμοστεί και να α, να ελεγχθεί. Αλλά να μην αφήσουμε α, κατά μέρος πάρα πολύ εύκολα τις επιδοτήσεις για την ανάπτυξη. Γιατί υπάρχει τέτοια, τέτοια σχετική πρόβλεψη α, στην ε, νομοθεσία για την προλόγηση θα πρέπει να συμπεριληφθεί λοιπόν το θέμα την, της χρέωσης και των χρεών και στο θέμα της φορολόγησης. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει με ενίσχυο τρόπο να αντιμετωπίζουμε και τα χρέη και τα equities. Και τέλος, υπομίζω τον τόκων, ουσιαστικά διαταράσσει τον φυσιολογικό τρόπο λειτουργίας των εταιριών που ουσιαστικά δανείζουν για να επενδύσουν. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώ. Και τέλο, κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω. Βλέπω ότι υπάρχει μια, ένα διστασμό για την προσμείωση. Tax credit αναφέρει ο Μάρκο Φέμπερ, η η Εύα Ζολή, στην 220 τροπολογία προσπαθεί να περιορίσει την απομείωση στα εργατικά έξοδα. Το καταλαβαίνουμε γιατί μία από τις ανησυχίες η οποία δεν είναι είναι ότι τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα και ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στις ε, δαπάνες ε, των, των εργαζομένων. Ε, μιας και πλησιάζουν τα επτά λεπτά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις τροπολογίες σας. Νομίζω ότι αποτυπώνουν ε, με πολύ ακριβή τρόπο και τις συζητήσεις που διεξαγάγονται στα εθνικά κοινοβούλια σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια, την κεφαλαγορά. Κάνουμε και επισκέψεις ε, σε διάφορες χώρες, περιοδία. Ε, τα πάμε και στην Ρουμανία και στην Ιρλανδία μας έχουν προσκαλέσει όλους παραδόξους. θεωρώ ότι αυτά θα επηρεάσουν και τις συζητήσεις στο Συμβούλιο προκειμένου να δούμε ποιο θα είναι το μελλοντικό ε, πρότυπο για την κοινή βάση φορολογίας εταιρεών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος. Τώρα, ο εισηγητή για την κοινή ενωπημένη βάση φορολογία εταιρεών, ο κ. Λαμασούρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και ο Πολ, δουλεύουμε εδώ και πολλές εβδομάδε. σε στενή συνεργασία προκειμένου να καλύψουμε όσο περισσότερες ανησυχίες έχουν τα εθνικά κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις. Ε, αναφέρθηκε το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα επισκέψεών μας και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι κατέθεσαν πολλοί άριθμες τροπολογίες και να υπενθυμίσω ότι για αυτό το φορολογικό θέμα του οποίου η σημασία υπενθυμίζεται από διάφορα πράγματα που βλέπουμε στον τύπο, στην επικαιρότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα αυτό το πλαίσιο δυστυχώ δεν μπορεί να συμμετάσχει στη λήψη των αποφάσεων. Απλώ νομοθετούμε. Και ξέρουμε ότι το Συμβούλιο Υπουργών δεν λαμβάνει πάντα υπόψη τι απόψει του Κοινοβουλίου για θέματα τέτοιου τύπου. Ο πολιτικός μας στόχος είναι να πετύχουμε το Συμβούλιο Υπουργών να υποχρεούται να αντιμετωπίζει επί της ουσίας διάφορα ουσιαστικά θέματα, να εξετάζει επί της ουσίας διάφορα ουσιαστικά θέματα που θέτει το διπλό αυτό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν τρεις στόχοι επί των οποίων ε, που, τους οποίους τονίζουμε. Μέσω της ε, κοινή ε, ενωπημένης βάσης πρέπει να βάλουμε τέλος στο φορολογικό μας πόλεμο. Μιλάμε για φορολογικό ανταγωνισμό. Στην πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια έχει μετασχηματιστεί σε πραγματικό πόλεμο. Κάποια κράτη-μέλη ουσιαστικά ε, κλέβουν τη φορολογική ας πούμε, βάση των άλλων κρατών μελών. Έγιναν πολλέ προτάσει λοιπόν και στον ΩΣΑ και αλλού για να σταματήσει αυτό ο πόλεμο. Δεύτερο στόχο. Να εναρμονίσουμε τον ορισμό τη ε, φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εναρμόνιση με σκοπό να εναρμονίσουμε. Έτσι. Ο, είναι αυτό ο σκοπός η εναρμόνιση και το δέχονται τα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δέχτηκαν μάλλον τα 15 κράτη-μέλη πριν από 20 χρόνια και έκτοτε εντάξει το ξεχάσαμε λιγάκι. Θέλουμε να έχουμε ένα φορολογικό χώρο ενιαίο μέσα στο, στο ενιαίο οικονομικό και δημοσιονομικό χώρο για όλες τις εταιρείες που δουλεύουν μέσα σε αυτόν τον ενιαίο χώρο. Τρίτον, να υποφελθούμε της ευκαιρίας για να εξυγχρονίσουμε και να πλουστεύσουμε την φορολόγηση των επιχειρήσεων στις χώρες μας. Αυτό ακριβώς κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και όταν λέω εξυγχρονίζουμε, προφανώς σημαίνει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το ειδικό πρόβλημα που θέτει η ψηφιακή οικονομία και οι ψηφιακές πλατφόρμες. Υπάρχουν διάφορες ιδέες που κυκλοφορούν και αναφέρθηκαν. Καταρχάς η πρωτοβουλία του, της γαλλικής κυβέρνησης, της σημερινής γαλλικής κυβέρνησης να υπάρξει με ένας έμεσος φόρος. Προτείνουμε για λόγους αποτελεσματικότητας και για να λάβουμε υπόψη τη σκοπιμότητα και τη σημασία που έχει αυτό το κείμενο να βάλουμε τη φορολόγηση των, φορολογικών, των ψηφιακών συγγνώμη, πλατφορμών στην ενιαία, στην ενοποιημένη ε, φορολογική βάση. Αυτή είναι η τριστόχη λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε αντί να είναι υποχρεωτικό οι μεγάλες επιχειρήσεις για τις υποχρεώσεις, να είναι μάλλον το σύστημα υποχρεωτικό για τι μεγάλε επιχειρήσει και ε, προαιρετικό για τι μικρέ, να ισχύει για όλε. Γιατί έτσι είναι και υπάρχει και ίσως ε, ανταγωνισμός και επιπλέον ε, ζητάμε και μια γιγάντια προσπάθεια από τις φορολογικές ε, υπηρεσίε. Επίσης, τα δύο κείμενα θα πρέπει να εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ όταν βλέπετε τις πολυάριθμε πολυάριθμες Θα θέλουμε και τα τρία C να εφαρμοστούν του CCCTB, ενιαία ενωπημένη βάση δηλαδή. Επίση, η φορολόγηση σε ένα κρατό μέλο. να γίνεται με διάφορα κριτήρια, ε, λαμβάνοντας υπόψη που έχει δραστηριότητες μία ε, πολυεθνική. Επίσης, μπορεί, αν εφαρμοστεί το νέο σύστημα, να έχουν περισσότερα φορολογικά έσοδα κάποια κράτη-μέλη ε, και κάποιες απώλειες ε, κάποια άλλα. Θα πρέπει να μειωθούν σύν το χρόνο αυτές οι ανισότητες και επίσης είμαστε πολύ ευαίσθητοι στο πρόβλημα της συγκεκριμένης εφαρμογής σε ό,τι αφορά το εύλογο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή, την απαραίτητη ευελιξία. Μίλησα για μια φορολογική επανάσταση εγώ για τις φορολογικές διοικήσεις που είναι υπεύθυνε. Και μην ξεχνάτε ότι δεν έχουν την ίδια ποιότητα όλε οι εφορίε, όλε οι φορολογικέ αρχέ. Τα θέματα είναι περίπλοκα ε, και πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ, έτσι. Αυτή είναι η βάση. Και με βάση όλα αυτά, δέχτηκα κάποιε τροπολογίε και απέρριψα κάποιε άλλε. Ε, ειδικά οι τροπολογίε που αρνούνται τι βασικέ αρχέ τη οδηγία. Δεν τι δέχομαι. Ε, Παραδείγματο χάρη το προαιρετικό σύστημα κτλ. Ένα κομμάτι υποχρεωτικό και ένα προαιρετικό. Επίσης, για το κατόφλι. Εγώ δεν θέλω κανένα κατόφλι. Ή το σύστημα είναι καλό και τότε γιατί να εξαιρέσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή το σύστημα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και τότε γιατί να τιμωρήσουμε τις μεγάλες επιχειρήσει, επιχειρήσεις απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών. Ας πούμε. Είναι απλό ε, σύστημα και πρέπει να εφαρμοστεί. Επίσης, θέλω να υπάρξει μια καλύτερη πραγματογνωμοσύνη για τις πολυάριθμες τροπολογίες ό,τι αφορά τον ορισμό ενός ομίλου και τις σχέσεις τις ενδοομιλικές. Εντυπωσιάζομαι από το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοι προτείνουν πάρα πολύ τεχνικές τροπολογίες. Θα πρέπει να τις εξετάσουμε. Είμαι βεβαίως πολύ ανοιχτό. Επίσης είμαι ανοιχτό σε τροπολογίες που αφορούν την σύνθεση και τη στάθμιση του τύπου για την ε, κατανομή, τη γεωγραφική κατανομή δηλαδή της φορολογικής βάσης ενός ομίλου, εννοείται εδώ. Λοιπόν, για τη μεταχείριση, ε, την αντιμετώπιση μάλλον των διαφορετικών τύπων που πρότειναν οι διάφοροι συνάδελφοι, πολύ ενδιαφέροντες όλοι αυτοί οι τύποι, όλες αυτές οι προτάσεις για τις τροπολογίες σε σχέση με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων ε, θα πρέπει να έχουμε αναλύσεις αντικτύπου βεβαίως για το μηχανισμό και τον ανάλυση του μηχανισμού αντιστάθμισης επίσης προφανώς θα πρέπει να γίνει Επίσης δεν έχω δυσκολία να δεχτώ τις τροπολογίες που υπενθυμίζουν ότι η τροπολογία παραμένει βασικά αρμοδιότητα των κρατών μελών Αυτά συνάδελφοι πρώτες αντιδράσεις εν θερμό σας ευχαριστώ όλους και όλες όσους ε, με τις τροπολογίες προσπαθήσατε να εμπλουτίσετε την έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο εισηγητές. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τους σκιώδους εισηγητές. Έχετε 7 λεπτά στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ κοιτάμε και τα εθνικά στοιχεία, η διαφορά μεταξύ των εγγράφων Παναμά και Paradise είναι, θεωρώ, ότι έχουμε πληροφορίες από άλλο πάροχο, αλλά ουσιαστικά οι πληροφορίες και οι μηχανισμοί είναι λίγο πολύ οι ίδιοι και έτσι σε ό,τι αφορά την ανάλυση του προβλήματος έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά σε αυτά τα οποία θα κοιτάξουμε και στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν ε, και άλλες ε, δημοσιεύσεις, γιατί φαντάζομαι ότι και από την, πέρα από τις εταιρείε που έχουν ήδη αναφερθεί και στην Φόντσεκα και την ε, εταιρεία αυτή τώρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία είναι κρεμή και τα οποία είναι ευαίσθητα. Αυτά έτσι προκαταρτικά. Να πω και κάποιες άλλες να καπώ και κάποια άλλα στοιχεία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια πρόταση για μια ένα συντελεστή ε, αξιολόγησης και προσμέτρησης ε, βάση φορολογίας ε, και επίσης τίθεται και το θέμα της κοινή ενοποιημένης βάσης. Αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε και αγαπητέ Πόλα, στο είπα και προσωπικά, ως Κοινοβούλιο θεωρώ ότι θα πρέπει να προτείνουμε ενιαία φορολογική βάση και φορολογικό συντελεστή. Δεν θα πρόκειται να ενθουσιαστεί φυσικά το, το Συμβούλιο γιατί δεν έχουμε άλλωστε και αρμοδιότητα στα θέματα φορολογικά, άρα θα πρέπει να δράσουμε με μεγάλη σύνεση και προσοχή. Αυτό το λέω έτσι εξ αρχής. Ε, αντιμετωπίζουμε υλικά μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι οι συνέπειε, ποιε θα είναι οι συνέπειε για τα φορολογικά έσοδα. Προσπάθησα σε εθνικό επίπεδο να συλλέξω σχετικέ πληροφορίε για το ποιο θα είναι τελικά το αποτέλεσμα ε, σε εθνικό επίπεδο για τα φορολογικά έσοδα, αλλά η κατάσταση φαίνεται είναι πάρα πολύ ασαφή. Και αυτό αποτελεί τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στην παρούσα φάση. Και επειδή υπάρχει ακριβώ αυτή η αβεβαιότητα, πιστεύω ότι θα πρέπει να δράσουμε μάλλον πιο προσεκτικά και διστακτικά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δύο μεγάλα κενά τα οποία υπάρχουν και αναφέρονται εδώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα ε, προσμείωση, σε ό,τι αφορά ε, την έρευνα και την ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Να σας πω σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της έρευνα και την καινοτομία. Εμείς πληρούμε τον ε, στόχο του 3% χωρίς να υπάρχει καν ε, δυνατότητα προσμείωσης ε, των φορολογικών υποχρεώσεων. Δεν μπορούμε λοιπόν να επενδύσουμε και παραπάνω στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Είμαστε σε ριακό σημείο. Υπάρχει μια άλλη χώρα δυτικά της Γερμανίας που έχει εισαγάγει τέτοια δυνατότητα φορολογικής προσμείωσης, απομείωσης. Υπάρχουν ε, άλλοι μηχανισμοί φυσικά πέρα από το μηχανισμό αυτό με τον οποίο μπορούμε να προωθήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ένα πιστοτικό σημείο μας σε ό,τι αφορά την φορολόγηση ιδιαίτερα για μικρές επιχειρήσεις και για νεαρές επιχειρήσεις που ενδεχομένως να μην έχουν ήδη πολλά κέρδη και σε τελική ανάλυση αυτοί που ωφελούνται από την μείωση της φορολογίας είναι οι μεγάλες ε, επιχειρήσεις, οι μεγάλες εταιρείε. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι μικρές εταιρείες, οι καινούργιες εταιρείες έχουν ε, ζημία γιατί πρέπει να καθιερωθούν στην αγορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τις επένδυσεις, το σχετικό σημείο. Φυσικά θέλουμε να προωθήσουμε τις κεφαλαίες Τώρα πώς θα γίνει αυτό με την φορολογία και το φορολογικό δίκαιο δεν είναι σαφές. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω κατά πόσο πραγματικά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί σωστό μέσο σε ό,τι αφορά την υπομείωση των τόκων, περαιτέρω Εγώ έχω καταθέσει σχετικές τροπολογίες. Αυτό θεωρώ ότι θα αυξήσει αυτό την ελκυστικότητα των κεφαλαίων χωρίς να υπάρχουν οι παραπλευρές απώλειες. Το θέμα της ψηφιακής οικονομίας μας απασχολεί όλους. Αλλά θα ήθελα να κάνω εδώ πέρα μια υποσημείωση, αγαπητέ Πρόεδρε. Στα πλαίσια της επισκεψής μας στο, στην Ουάσιγκτον ε, στην, ε, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είχα, είχε προβλεφτεί και επίσκεψη ε, με τον ε, επικεφαλής του Διεθνούς Ταμείου η οποία κυρώθηκε τελευταία στιγμή. Είναι πάρα πολύ κρίμα και φυσικά το θέμα της ψηφιακής οικονομίας αποτέλεσε σημαντικό θέμα στο οποίο μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε και πρέπει ασφαλώς να κοιτάξουμε κατά πόσον διεθνώς πώς υπάρχει συντονισμό σε ό,τι αφορά τον ορισμό της ψηφιακής έντρας εταιριών. Φυσικά, όσα θέλει να κοιτάξουμε το θέμα αυτό, ενδεχομένως να πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση αυτή για να μπορέσουμε να καλέσουμε και τον ΩΣΑ στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή του Κοινοβουλίου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει συντονισμό. Υπάρχουν διάφορε πρωτοβουλίε από διάφορα κράτη-μέλη για το πώς ε, θα γίνει ή θα μπορούσε να γίνει ε, φορολόγηση του κύκλου εργασίων. Αν είναι δύσκολο να φορολογήσουμε τα κέρδη, πώς θα το κάνουμε αυτό, θα το σκεφτούμε βέβαια. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν δρόμο προκειμένου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρούμε έναν ορισμό για την ε, εικονική έδρα ε, εταιριών και το πώς θα μπορούσαμε να, να συγχρονιστούμε και να συντονιστούμε με τον ΩΣΑ. Γιατί θεωρώ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να ηγηθούμε τη όλη διαδικασία, γιατί αυτό αποτελεί ένα από τα μεγάλα εκκρεμή ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμίσουμε. Θα πρέπει να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε λοιπόν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η πρώτη και η καλύτερη, αν θέλετε, στη διαδικασία αυτή και προκειμένου να συγχρονιστεί με τις δράσεις μας και όσα. Ε, σε αυτά θα περιοριστώ και θα ήθελα να πω ότι ανυπομονώ για τη μελλοντική συνεργασία. Ελπίζω στη τελική ανάλυση να βρούμε έναν ισορροπημένο συμβιβασμό που θα μας ε, δώσει δυνατότητες να συνεχίσουμε και τις διαπραγματεύσεις στους κόλπους του Συμβουλίου. Γιατί αυτό να σας με απασχόλει πάρα πολύ. Τι να την κάνουμε τη σούπερ λύση άμα την βρούμε, αν δεν την δεχτεί το Συμβούλιο. Αν θέλουμε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουμε, να είμαστε ρεαλιστές στις προτάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you um, very much. Ευχαριστώ. Ουγκμπαγή από τους Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και ο συνάδελφος, δεν έχω την αίσθηση ότι τυχαία γίνεται αυτό το σήμερα. Σήμερα μιλάμε για την ε, σύγκληση ε, για να έχουμε μια οικονομική πολιτική πιο στονισμένη και να καταπολεμήσουμε την ε, φορολογική, τη φοροδιαφυγή. Επίσης, τα Paradise Paper μας υπενθύμησαν ε, ε, τους φορολογικούς παραδείσους, έχουμε και τα Lux ε, Leaks και τα λοιπά. Εδώ αυτά τα papers μας έδειξαν τις ε, ε αθέμητες φορολογικές πρακτικές ή τις ε, παράνομες φορολογικές πρακτικές. Μία ενοποιημένη φορολογική βάση νομίζω ότι θα μας επέτρεπε να εξασφαλίσουμε ότι φορολογούμε την, τα κέρδη εκεί που δημιουργείται η οικονομική αξία. Το τα κείμενα των δύο εισηγητών αποτελούν μια πολύ καλή ε, βάση εργασίας. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ε, πάρα πολλά πράγματα υπόθηκαν. Ε, θα ήθελα να κάνω απλώς κάποιες παρατηρήσεις για τις διάφορες τροπολογίες. Πρώτη παρατήρηση, ε, Κρίμα για τη στάση κάποιων μελών αυτής της Επιτροπής που, ζουν, που ζητούν απλώς να απορρίψουμε την οδηγία. Νομίζω ότι όλοι οι παράγοντες της κοινωνίας συμφωνούν ότι αυτή η οδηγία είναι εκ των ονουκάνευ, ε, απλουστεύει τη ζωή των ε, επιχειρήσεων, ε, που φορολογούνται σε διάφορε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και είμαστε και πιο αποτελεσματικοί κατά των φορολογικών απατών. Ε, δεν θέλω λοιπόν ε, αυτέ τι τροπολογίε που απορρίπτουν απλώ την οδηγία. Χαίρομαι που πολλοί ευρωβουλευτέ θέλουν να αντιμετωπίσουμε από κοινού τι διεκθέσει, γιατί αν θέλουμε πραγματικά η πρόσβαση να είναι αποτελεσματική και να αλλάξουν τα δεδομένα, πρέπει να ε, το να έχουμε μία κοινή βάση φορολογία χωρί ενοποίηση δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Ε, τα δύο πράγματα είναι αλληλένδετα νομίζω. Επίση, κάποιο συνάδελφο το είπε, αλλά το τονίζω και εγώ, ε, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τι φορολογικέ προκλήσει ε, που δημιουργεί, η ψηφιακή οικονομία, να εξυγχρονίσουμε την ε, φορολόγηση στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας καλύτερα τη μεγάλη κινητικότητα των κεφαλαίων, το είπαν διάφοροι συνάδελφοι, Τέταρτη παρατήρηση. Τους μηχανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε σε αυτή την πρόταση το μηχανισμό με σκοπό να προωθήσει τις επενδύσεις για την καινοτομία, το υποστηρίζουμε, και από την άλλη να προωθήσει την χρηματοδότηση μέσω της χρέωσης, ε, μέσω της λαμβάνοντα υπόψη τις, ε, τα περιουσιακά στοιχεία. Ε, εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα για τις δύο επιχειρήσεις. Ε, δεν θα πρέπει εδώ να δημιουργήσουμε νέα κενά, ενώ ο στόχος μας είναι να καλύψουμε ας πούμε, τα κενά που υπάρχουν τώρα. Επίσης θα πρέπει να προοδεύσουμε στη συζήτηση για τα βασικά στοιχεία που είναι ο φορολογικός συντελεστής και το κατόφλι από το οποίο η, μια επιχείρηση εντάσσεται στην οδηγία ή όχι. Εμείς ως σοσιαλιστές θεωρούμε ότι όλες οι πολυεθνικές θα πρέπει να εντάσσονται στην οδηγία αυτή, σε αυτό το κείμενο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε διάκριση, δηλαδή ανάλογα με το τζίρο, με τον κύκλο εργασιών, δεν υπάρχει λόγος, γιατί ε, να διαρρέσουμε δηλαδή εμείς τις πολυεθνικές μα αντί να τι αντιμετωπίσουμε ισότιμα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι και αξιόπιστη αλλά και αποτελεσματική ε, και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να επιλύσει αυτό το βασικό πρόβλημα. Είμαστε όλοι εκλεγμένοι και όλοι λογοδοτούμε. Κανένας δεν μπορεί εδώ να εξηγήσει στους πολίτες ότι ένας φορολογικός τελεστής 0% ή ακόμα και 12,5% δεν έχει σαν βασικό στόχο, αν όχι μοναδικό, να αφαιρέσει φορολογικά έσοδα ας πούμε, από τη μια χώρα και να τα πάει σε μια άλλη. Τρελαθούμε. Ε, επίσης, ε, μια επιχείρηση που έχει 500 εκατομμύρια ε, κύκλο εργασιών, πώς μπορεί να παίζει με τις αναντιστοιχίες και τις διαφορές που έχουν 28 χώρε μα, τα 28 φορολογικά μα συστήματα. Γι' αυτό θέλουμε ένα πραγματικό φορολογικό συντελεστή 18% για όλε τι επιχειρήσει μηδενιά εξαιρουμένη. Επίση, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το, για το πλαίσιο μέσα στο οποίο η πρόταση αυτή θα πρέπει να συζητηθεί ε, και εδώ αλλά και στο Συμβούλιο. Μην ξεχνάτε ότι η πρόταση του 2011 ε, απέτυχε στο Συμβούλιο και 28 κυβερνήσει δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν και να υπάρξει ομοφωνία που απαιτείται για φορολογικά θέματα. Από τότε η επικαιρότητα μα δείχνει ποιε είναι οι συνέπειε αυτή τη αποτυχία του Συμβουλίου. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό το κείμενο θα μπορέσει να καταλήξει με μια μαζική στήριξη στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα ακόμα μια φορά να χαιρετήσω τη δουλειά που έκαναν οι δύο εισηγητέ και να του ε, ευχηθώ ε, να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη ε, θέση του Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να πιέσουμε και το Συμβούλιο για να συμφωνήσει προ αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά, Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο Σάντερ Λούνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Χιούγκ έχει ε, δίκιο. Συνεχίζω να πιστεύω ότι καλά κάναμε και απορρίψαμε αρκετές τροπολογίες ε, και σήμερα θα ήθελα να εξηγήσω για ποιους λόγους το κάναμε αυτό. Ο στόχος της κοινή βάσης φορολόγησης και της κοινή ενοποιημένης βάσης φορολόγησης είναι ε, θεμητός. Υπάρχουν όμως και άλλα μέσα, πιο έξυπνα, πιο αναλογικά. Νομίζω λοιπόν ότι το CCTB αποτελεί υπερβολικό περιορισμό για τα κράτη-μέλη που ε, εμποδίζει τα κράτη να είναι δημοσιονομικά ανταγωνιστικά και κάτι τέτοιο θα επηρεάσει αρνητικά ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανταγωνιστικότητά της. Ε, αυτό είναι που ε, μας κάνει πιο δυνατούς η ανταγωνιστικότητα. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δίκαιο οι πολυεθνικές να μπορούν να χρησιμοποιούν το ε, επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό για να μειώνουν ε, τις φορολογικές οφειλές τους σε σύγκριση με μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τα μέσα να προβούν σε τέτοιο φορολογικό σχεδιασμό. Συμφωνούμε ότι πρέπει να πληρώνονται φόροι εκεί που δημιουργούνται τα κέρδη και αυτός είναι ο, ο λόγος που έχουμε δρομολογήσει δέσμες ε, μέτρων σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να γίνουν τα φορολογικά συστήματα πιο διαφανή και πιο απλά. Έχουμε λάβει υπόψη και την πρωτοβουλία BEPS του ΟΣΑ τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τις ε, σχετικές ε, συστάσεις. Έχουμε συμφωνήσει ότι η εφαρμογή κάποιων προτάσεων του ΟΣΑ που επηρεάζουν άμεσα την εσωτερική αγορά έχουν θετικό αντίκτυπο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι έχουμε ακόμα δρόμο, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τον επιμερισμό των φορολογικών κερδών. Τώρα κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να ορίσει το δικό του εταιρικό φόρο. Είναι ξεκάθαρη έκθεση του εισηγητή ΤΑΝΚ. Σήμερα υπάρχει το περιθώριο να ε, επιδίδονται τα κράτη-μέλη σε έναν φορολογικό ανταγωνισμό το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει ένας ελάχιστος φορολογικός συντελεστής. Ξέρω ότι κάποιοι ονειρεύονται υψηλότερους φόρους ε, για τις πολυεθνικές. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ενισχύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι το όριο όμως τι ε, μας επιφυλάσσει το μέλλον. Στη συνέχεια για τι πράγμα θα συζητήσουμε, για περιβαλλοντικούς φόρους, για φόρο εισοδήματος κτλ. κτλ. Αυτή η πρόταση έχει στόχο την εναρμόνιση των φορολογικών πολιτικών σε ε, ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να ενισχύσουμε την ε, ενιαία αγορά. Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός είναι ε, θετικός και πρέπει να τον ενθαρρύνουμε. Ο Μισελ Οζόν, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στο, ε, στην δρομολόγηση των δημοσιονομικών σχέδιων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ότι υπάρχει τόσο πολύ φορολογικός ε, σχεδιασμός, ε, φορολογικός ανταγωνισμός. Και η μεγάλη τραγωδία είναι ότι οι φορολογικοί συντελεστές έχουν πέσει από το 36% στο 22%. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι καλό. Είναι καλό για την οικονομία, για τις επενδύσεις, για τους επιχειρηματίες και για τους καταναλωτές. Και αν κοιτάξουμε περαιτέρω το θέμα του ανταγωνισμού, εντός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, σήμερα αν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος από τη φορολογική νομοθεσία πολύ απλά πηγαίνει σε μια άλλη χώρα. Ε, αυτό έχει συμβεί πολλές φορές. Κάποιοι έχουν φύγει από τη Γαλλία. Γάλλοι έχουν μεταφέρει την έδρα τους στο Λονδίνο. Και ε, στο Λονδίνο πλέον υπάρχουν περισσότεροι ε, Γάλλοι επιχειρηματίες από ότι στο Στρασβούργο. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μακρόν ε, προχωρεί πολύ λογικά γιατί ο φορολογικός εντελεστής θα κάνει την Γαλλία πιο ανταγωνιστική και αυτό θα θέσει την Γαλλία επίσης όρις με άλλα κράτη-μέλη. Σε κάποιους δεν αρέσει αυτός ο φορολογικός ανταγωνισμό. Προτιμούν έναν φορολογικό πόλεμο, όμως εγώ δεν συμφωνώ. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο όμως είναι η απώλεια κυριαρχία θα πλήξει κυρίως τα μικρότερα κράτη μέλη, όπως η δικιά μου χώρα, το Βέλγιο, αλλά και τις κατώ χώρες, στην ε, Ιρλανδία, θα πληγούν όταν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, γιατί τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη έχουν ήδη οικονομίες κλίμακας, έχουν ήδη αναπτυγμένες οικονομίες, έχουν ευκαιρίες που τα μικρότερα κράτη-μέλη δεν έχουν. Τα μικρότερα κράτη-μέλη πρέπει να φερθούν έξυπνα και πρέπει ε, να έχουν ελκυστική φορολογική νομοθεσία. Χρειαζόμαστε λοιπόν έξυπνη δημοσιονομική πολιτική προκειμένου να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Τέλος, δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε το CCTB και το CCCTB. Χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα για να καταπολεμήσουμε τις δράσεις ε, των φορολογικό, επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό των ε, πολυεθνικών γιατί στο παρελθόν κάποιοι ε, έκαναν επιλογές εγκαταλείποντας ένα κράτος μέλους προς όφελος ενός άλλου κράτος μέλους αλλά ο κίνδυνος των μέλων είναι να φύγουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εξηγήσουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την Ευρώπη αν οθήσουμε τις εταιρείες να φύγουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και πολύ φοβάμαι ότι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το να μετακινηθούν σε μια άλλη φορολογική δικαιοδοσία είναι πάρα πολύ α, περίπλοκο. Είναι σχεδόν αδύνατο, ναι, αλλά θα του δώσει... Σχόλια εκτό μικροφώνου. Okay, Ναι, θα του δώσετε συμβουλέ. ε. αδιαφυσβήτητα. Μάλιστα. Από την ομάδα τη Άλντε. Ο κύριος Γεζέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι τι θα κάνει ο κόσμος και πώς θα ψηφίσει τον θα λάβει χώρα και τον Brexit. Ε, εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστήσω τους εισηγητές για τη δουλειά που έχουν κάνει για το θέμα αυτό, για το φάκελο αυτό. Να σας υπενθυμίσω εκ νέου τη σημασία των δύο προτάσεων για την ενίσχυση της ε, ενιαίας αγοράς και για τη μεταρρύθμιση των προλογικών συστημάτων. Επίσης, η Επιτροπή μα έχει λάβει χώρα, έχει λάβει υπόψη ναι, και τα έγγραφα του Παναμά και τα έγγραφα Paradise. Όλα αυτά καταδεικνύουν πόσο απαραίτητο είναι να αντιμετωπιστεί ο επιθετικός φορολογικός ε, σχεδιασμός. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε τις πρακτικές αυτές. Αλλά αυτό λείπει από την πρόταση. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη χρειάζονται στις πρωτοβουλίες αυτές. Το έχω κάνει άλλωστε αυτό στις τροπολογίες μου. Επειδή όμως πολύ πιθανόν σε τελική ανάλυση αυτή η ενοποίηση να αποτελέσει τμήμα μόνο του δεύτερου της δεύτερης φάσης του συστήματος υπάρχει και ανάγκη να υπάρξει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για την επίλυση των διαφορών γιατί αυτός ο μηχανισμός δεν θα είναι και υποχρεωτικός για όλες τις εταιρείες κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό στο οποίο επίσης αναφέραμε στις τροπολογίες μου είναι η φορολόγηση του ψηφιακού κλάδου. Θα πρέπει να ορίσουμε εκ νέου το, μόνιμο κατάστημα για να συμπεριληφθεί και αυτή η ψηφιακή τη μόνιμη εγκατάσταση για να λάβει, ληφθεί υπόψη και η ψηφιακή διάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή η δικαιοδοσία ορίζεται μόνο με τη φυσική παρουσία της εταιρείας. Μετά την τελευταία ανταλλαγή απόψεων. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ε, επικίνδυνο να, να ξεκινήσει εδώ η συζήτηση του ελάχιστου συντελεστή, ξέροντα και ποιε είναι οι θέσει των κρατών μελών. Γιατί αυτό θα δώσουν πιο πολύ λόγο να αντιδράσουν τα κράτη-μέλη. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το θέμα δεν είναι η εναρμόνιση του φορολογικού συντελεστή. Αν θέλουμε πραγματικά να λειτουργήσει το σύστημα και η ομάδα μου κατέθεσε κάποιε σχετικέ τροπολογίε. Επίσης, κάναμε τροπολογίες για τις διατάξεις ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών επιφορολογικών ζητημάτων. Πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό για την ομάδα μου. Τέλος, καταθέσαμε τροπολογίες ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή και τη συμπερίληψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει αξιολόγηση του αντικτύπου του εθελοντικού, εθελούσιου χαρακτήρα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να ζυγίσουμε πλανεκτήματα και μειονεκτήματα για να καταστεί ή όχι υποχρεωτικό το σύστημα για τις μικρομεσαίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ζολή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την αρχή της ετίας ε, του Κοινοβουλίου γίναμε μάρτυρε τριών μεγάλων σκανδάλων ε, που αφορούν, ε, που αφορούν ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις. Και όλοι οι εθνικιστές τους απαντούν ή μάλλον καλό θα ήταν να τους απαντήσουμε ότι καταλάβαμε το πρόβλημα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί τώρα την κατάλληλη νομοθεσία, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του να μην πληρώνουν πουθενά φόρο οι πολυεθνικές. Και πώς το αντιμετωπίσουμε μέσω του CCTB. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι οι δύο αυτές οδηγίες να εξεταστούν παράλληλα. Γιατί φοβάμαι ότι αν περιοριστούμε μόνο στην πρώτη, στην κοινή βάση φορολογία εταιριών, η δεύτερη για την κοινή δοτημένη βάση φορολογία, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Λαμβάνοντα υπόψη το, τις προσδοκίες της κοινή γνώμη και τον αριθμό των σκανδάλων, λογικό είναι να θέλουμε να τεθούν παράλληλα αυτές οι δύο οδηγίες σε ισχύ ε, το 2020, όπως λέει και οι συγκητές μας. Οι προσδοκίες που υπάρχουν ε, έρχονται σε αντίθεση με τους φόβους που προκάλεσε το προηγούμενο μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο από την προηγούμενη ε, απόπειρα. Γιατί χρειάζεται ομοφωνία και ξέρετε πολύ καλά ότι το Λουξεμβούργο ούτε η Ιρλανδία θέλουν να υποστηρίξουν και το ΕΒ θέλουν να υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο. Επομένως, Κομισιόν, σας καλούμε να, να χρησιμοποιήσετε το άρθρο 116 να το ε, να το επικαλεστείτε και να θεωρήσετε ότι πρόκειται για μία ε, στρέβλωση, του ανταγωνισμού. Και να περάσετε στην εξέταση, δηλαδή με απλή πλειοψηφία. Επίσης, να περάσετε στην ενισχυμένη συνεργασία με τη δυνατότητα τελικά για αυτούς που συνεργάζονται να καταγγέλουν τις διμερείς φορολογικές συμφωνίες με τα κράτη δηλαδή που δεν παίζουν και αυτά ε, με δίκαιους όρους, ούτως ώστε να τα πιέσουμε και να μην, για να μην δέχονται πλέον ε, προϊόντα, ας πούμε, έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, για τη φορολογητέα βάση ε, έχω υποβάλει τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας το επίπεδο φορολόγησης, γιατί αλλιώς θα περάσουμε από, την, από τον ανταγωνισμό για τη φορολογική βάση στην, στον ανταγωνισμό για τους τελεστές. Εγώ προτείνω να στελεστεί στο ύψος του 20% και ένα τμήμα αυτού να πηγαίνει στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ένα τμήμα από τα έσοδα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να φορολογούμε την ψηφιακή οικονομία. Όλοι γνωρίζουμε την σημερινή κατάσταση όπου είναι δυνατόν. Φερρυπίν, η Google στη Γαλλία να έχει 700 ε, άτομα, ε, χιλιάδες ε, υπολογιστές και να, και να έχει δεν ξέρω πόσα γραφεία, ας πούμε, τετραγωνικά μέτρα ολόκληρα, ας και να λέει «Α, δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση». Ε, να την ορίσουμε τη μόνιμη εγκατάσταση και να υπάρχει και η έννοια της ιονή μόνιμης εγκατάστασης. Και θα πρέπει επίσης στον τρόπο αναδιανομής των κερδών να έχουμε κριτήρια, ούτως ώστε να λάβουν υπόψη το business model το επιχειρηματικό μοντέλο της ψηφιακής οικονομίας. Δηλαδή τα έσοδα που δημιουργούνται από την ε, συλλογή πληροφοριών ή από τον αριθμό των χρηστών σε μια πλατφόρμα ας πούμε, ψηφιακή. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητήσουμε και είμαι πεπισμένη ότι θα βρούμε συμβιβασμού για το θέμα αυτό. Έξυπνου συμβιβασμού που να λειτουργούν στην πράξη. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα του debt bias, ε, δηλαδή της τρέβλωσης λόγω χρέους, ε, του σημείου αυτού που πρότεινε η Κομισιόν, νομίζω ότι η λύση της ε, Κομισιόν δεν είναι καλύτερη. Να επιτρέψουμε δηλαδή τα, τους τόκους ας πούμε, μάλλον τις, αυτή την λογική που υπάρχει στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή, να περιορίσουμε τη διάρκεια του χρόνου απομείωσης ε, των ε, χρεών, δηλαδή αφαίρεσης των χρεών. Υπάρχουν διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν ε, γίνει για το θέμα αυτό. Βλέπετε ότι υπάρχουν εταιρείε που επί 15 χρόνια δεν έχουν πλώσει φόρο. Γιατί έχουμε αυτή την χρέωση, ας πούμε, η οποία μεταφέρεται από χρόνο σε χρόνο. Ιστοδυνικές όπως σε ό,τι αφορά ε, την έκπτωση του κόστους ε, για την έρευνα και καινοτομία, ε, θα πρέπει να εξαιρέσουμε το χρηματοπιστωτικό τομέα, ούτως ώστε να πληρώνει ο φορολογούμενος για τοξικά προϊόντα, ας πούμε. Αντίθετα, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε φυσικά την καινοτομία με επιχορηγήσεις και με εγγύηση, των, με εγγυημένα δάνεια, του οποίου εγγυητής θα είναι το κράτος. Πιστεύω ότι θα βρούμε πολύ καλές συμβαστικές λύσεις με τους εισηγητές, γιατί μας πιέζει η επικαιρότητα και είναι κατεπίγουσα η κατάσταση. Δεν μπορούμε να, κρατήσουμε, να δεχτούμε να διαιωνίζεται μια τέτοια κατάσταση. Βλέπετε τα σχόλια που υπάρχουν στα Panama Papers. Ότι όλα αυτά, όλε αυτέ τις πρακτικές είναι νόμιμες. Ε, όχι, δεν πρέπει να είναι πια νόμιμες. Ο, προ, ο επόμενος, ο Μάρκο Βάλλη, είναι ο επόμενο ε, εισηγητή. Ευχαριστώ. Όπως διάφοροι συνάδελφοι έχουν ήδη πει, προείπει, και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι μετά το σκάνδαλο των Paradise Paper που έβγαλαν στη φόρα τα πάντα paper, είναι σημαντικό να προωθήσουμε πολύ πιο γρήγορα αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί όλοι τα έχουμε μπροστά στα μάτια μας αυτά τα θέματα που συνιστούν πραγματικά φορολογική έλλειψη δικαιοσύνης. Μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, ας πούμε θα πρέπει προφανώ όλα τα θεσμικά επίπεδα να δράσουμε ταχύτητα. σω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μα δώσει ένα κατάλογο το συντομότερο δυνατό, γρήγορα, ε, το συντομότερο δυνατό, συγγνώμη, ένα κατάλογο με χώρε που δεν συνεργάζονται. Ή χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, χρησιμοποιούν πρακτικέ αθέμητε απέναντι στο σύνολο. Επίση, για τι προτάσει. Μα αρέσει η πρόταση και η προσπάθεια που κάνανε οι σκιώδεις εισηγητές, ειδικά για να ενισχυθούν οι κανόνες για το CCCTB και να κλείσουν τα παραθυράκια και όλες τις δυνατότητε για διαιτησία. Πρώτο σημείο που θα ήθελα να πω. Η πρόταση που θεωρούμε ότι είναι σημαντική δεν εγγυάται μια πραγματική ενοποίηση. Γιατί υπάρχουν κάποιες ασυμμετρίες που παραμένουν σε επίπεδο λογιστικό και σε επίπεδο εθνικό. Είναι λοιπόν σημαντικό να προτείνουμε ότι ένα χρόνο μετά από την, από την ε, εισαγωγή των ε, οδηγιών αυτών να υπάρξει μια άλλη πρόταση, ένα χρόνο μετά έτσι, η θέση ισχύει, να υπάρξει μια άλλη πρόταση, ούτως ώστε να υπολογίσουμε καλύτερα τον, ε, την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας, ούτως ώστε να μην υπάρχουν οι ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, το πακέτο θα πρέπει να εισαχθεί, δηλαδή δύο οδηγίες παράλληλα να τεθούν σε ισχύ. Γιατί αλλιώ, μπορεί να έχουμε καθυστερήσεις για τη δεύτερη πρόταση. Ε, είμαστε κατά επίσης μιας μεταβατικής ε, περίοδου και να αντισταθμίσουμε τις ε, ζημίες ας πούμε των θυγατρικών είναι αντιπαραγωγικό. Τώρα για το κατόφλι εμείς προτείνουμε ένα κατόφλι 50.000 Συγγνώμη, 50 εκατομμύρια. 50 ε, ε, οι εταιρείε που έχουν ε, τζίρο κάτω από 50 εκατομμύρια δεν εντάσσονται στην πρόταση για να μην τι πλήξουμε. Ειδικά σε εταιρείε οι οποίε δραστηριοποιούνται μόνο στο, σε εθνικό επίπεδο. 50 εκατομμύρια είναι το κατόφλι, το οποίο θα συμμετέχει, θα λάβει υπόψη σχεδόν όλε τι τις πολυεθνικέ εταιρείε δεν θα βγάλουμε απ' έξω τις πολυεθνικές εταιρείες, ενώ θα γλιτώσουν διάφορες μικρομεσαίες που δραστηριοποιούνται ειδικά σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, όλες οι εμπορικές ε, επιχειρήσεις, ακόμη και αυτές που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία, να φορολογούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο αυτές που έχουν ε, μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση. Επίσης, είναι σημαντικό ε, να μειωθούν υπερβολικές εκπτώσεις, και τα κτλ. Γιατί δημιουργούνται τεράστια προβλήματα ε, με τα κτλ. Όλα αυτά τα προβλήματα που τα έχουμε συζητήσει, ας πούμε. Ειδικά στην Επιτροπή Τάξη, ας πούμε. Τα Panama Papers, είδατε τι προβλήματα δημιουργούνται εκεί με τις απομειώσεις. Ε, επίσης, οι επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα. Γιατί αλλιώς ε, δημιουργούνται διάφορα παραθυράκια ε, τα οποία εκμεταλλεύονται οι πολυεθνικές λόγω αυτού του μέτρου που υπάρχει για την έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία. Τώρα για τις τρίτες χώρες, τι προτείνουμε. Το πρόβλημα της ε, μεταφοράς κερδών προς αυτές τις χώρες είναι πολύ σημαντικό. όχι, να μην φορολογούμε μόνο το παθητικό της των επιχειρήσεων. Επίσης, για τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, η Κομισιόν θα πρέπει να προωθήσει μια νέα νομοθετική πρόταση και, και οποιαδήποτε πρόταση κάνει για τον φορολογικό συντελεστή θα πρέπει να βασιστεί σε μια μελέτη συγκριτική Επίση, οι σκιώδει έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Είδα τι ε, τροπολογίε τη ε, Γκουε και των Πράσινων, μου άρεσαν, αλλά και οι υπόλοιπε τροπολογίε σε καλό δρόμο είναι. Επομένω, νομίζω ότι μπορεί να βγει μια καλή δουλειά, ένα καλό προϊόν από αυτό το Κοινοβούλιο για να κλείσουν τα παραθυράκια. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ξαναδώσουμε το λόγο στον ε, ε σκιώδη εισηγητή της Άλντε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες σας. Τις εξέτασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να είναι ξεκάθαρο ε, ε όσους έχουν ακόμα αμφιβολίες ότι το CCTB και το CCCTB είναι οι μόνες λύσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη φορολόγηση των εταιριών. Αυτό δεν θα αφαιρέσει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ανταγωνιστούν το ένα το άλλο με φορολογικούς ε, συντελεστές. Κάτι τέτοιο πρέπει να παραμείνει δυνατό. Οποιαδήποτε πρόταση για ελάχιστο ή μέγιστο φορολογικό συντελεστή πρέπει να υποστηριχτεί από στοιχεία που ε, δείχνουν ότι δεν θα καταρρεύσει το σύστημα. Δεν πρέπει να επιδιώκουμε μόνο τη συνεχή μείωση των φορολογικών συντελεσών. Σε όσους φοβούνται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χάσει την ανταγωνιστικότητά της, απαντώ το εξής. Η δίκαιη φορολόγηση με αποτολισματικούς συντελεστές θα προσφέρουν νέο κίνητρο στα κράτη-μέλη για... και πιο ελκυστικά για επενδύσεις. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει πιο ελκυστική. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, συμφωνώ ότι πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών. Πρέπει να αναρωτηθούμε όμως αν αυτό θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους των ε, προτάσεων και δεν είμαι σίγουρη ότι θα το επιτύχουμε. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ίσως χρειαστούν κάποιες προσαρμογές, όμως αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί περαιτέρω ευελιξία προκειμένου να υπάρξει ευελιξία στο CCCTB δεν θα πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις. Κάτι τέτοιο θα είναι αναποτελεσματικό και δεν θα διασφαλίσει τη ε, διαφάνεια που επιδιώκει αυτή η πρόταση. Η μείωση του κατοφλού πρέπει να είναι αναλογική και πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο πρέπει να μειωθεί το κατόφλι προκειμένου να ε, ε, αυξηθεί επαρκώς η φορολογική βάση. Έτσι λοιπόν είμαι σίγουρη ότι θα επιτύχουμε συμφωνία. Σε αυτή την πρόταση όμως λείπουν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα μια βιώσιμη προστασία για τα κράτη-μέλη σε περίπτωση που δημιουργηθεί σημαντική απώλεια φορολογικών εσόδων. Δεύτερον, ένα σύστημα επίλυσης διαφορών ε, σε περίπτωση διαφορά ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Για το πρώτο πρόβλημα, ο εισηγητής προτείνει ένα ταμείο αποζημίωσης. Πιστεύω όμως ότι αυτό δεν θα ε, μας επιτρέψει να αντιμετωπίσει ε, ε, αποτελεσματικά το πρόβλημα. Και ρωτώ το εξής. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι απώλειες φορολογικών εσόδων θα οφείλονται μόνο στο CCCTB. Πώς θα το υπολογίσουμε αυτό δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τις διαφορές ανάμεσα σε κράτη-μέλη εξαιτίας της εφαρμογής των μαθηματικών τύπων. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να εφαρμοστεί ένα ε, ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα επίλυσης διαφορών. Για να γίνει πιο ισορροπημένος ο τύπος υπολογισμός και να εξυγχρονίσουμε το σύστημα είναι να βεβαιωθούμε ότι συμπεριλαμβάνονται οι ψηφιακές επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις της Κομισιόν. Χρειαζόμαστε όμως συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε βραχυπρόθεσμα. Όμως αλλάζοντας το μαθηματικό τύπο πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε νέα κενά. τέλο θα ήθελα να τονίσω ότι και τα δύο συστήματα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την απαραίτητη αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, uh, Ευχαριστώ. Τελειώσαμε λοιπόν ε, με τους σκιατές να περάσουμε στην διαδικασία Catch the Eye. Ο κ. Σόγκμαρκ έχει ζητήσει το λόγο. Και αν δεν θέλει κανείς άλλος, ο κύριος Χέις, αν θέλει κανείς άλλος, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο σημείο εκκίνηση να πω αυτά που αναφέρατε για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ένα πρόβλημα ότι οι νεοφυεί και οι εταιρείε νέα τεχνολογία φεύγουν στο εξωτερικό όταν είναι μικρέ, γιατί χρειάζονται πιο ευρεία κεφαλαία αγορά. Θα πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη, αλλά επίση χρειάζονται να δουν που έχουν τις καλύτερες ευκαιρίες να αναπτυχθούν. Και επίσης όταν μετακινούνται μεγάλες εταιρείε, αυτό επηρεάζει και τις μικρές εταιρείε, γιατί προφανώς είναι συμβιωτική η ύπαρξή τους και η ανάπτυξή τους. Εγώ από πλευρά μου και όπως το βλέπω, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μία σαφή παραβίαση της επικουρικότητας, η οποία και προκύπτει από τις ενστάσεις διάφορων εθνικών κοινοβουλίων. Η φορολογία είναι εθνική αρμοδιότητα. Καλωσορίζω το γεγονός ε, της αυξημένης, ενισχυμένης συνεργασίας στο πλαίσιο του ΩΣΑ, στο πλαίσιο άλλων διεθνών ε, οργανώσεων και πιστεύω ότι καλό είναι να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό διαφάνεια. Αλλά σε διάφορες περιπτώσεις ε, δεν θα πρέπει να μπαίνουμε στα, στις δικές ε. Και δεν είναι και απλό να γίνει αυτό, γιατί τα διαφορετικά αυτά φορολογικά συστήματα ουσιαστικά είναι έκφανση της διαφορετικής ε, ανάγκης που έχουν τα κράτη-μέλη για να χρηματοδοτήσει. Και αυτό συμβαίνει και σε δική μου περίπτωση. Κάποιοι έχουν χαμηλότερη και αυτοί που έχουν υψηλότερη φορολογία σε διάφορες περιπτώσεις έχουν πιο πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Και αυτό έχει την ε, ελκυστικότητά του. Αυτό πιστεύουμε. Οι καλύτερες υποδομές, οι καλύτερες χρηματοδοτήσεις σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη και αυτές ε, αποτελούν διαφορετικές ε, συνιστώσεις και διαφορετικούς παράγοντες. Αλλά τα κάτι μέλη έχουν και διαφορές οι διάφορε χώρε έχουν διαφορετική αγορά εργασία, διαφορετική βιομηχανία. Δεν υπάρχει μία ανία λύση. Και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούν λίγο καλύτερα οι εισηγητέ και οι συνεισηγητέ. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε διεθνέ επίπεδο, σε ψηφιακό επίπεδο. Η ψηφιακή οικονομία όμω δεν μπορεί να ακολουθήσει την παλιά βιομηχανική λογική. Ποια είναι λοιπόν η αξία. Στην Καλιφόρνια, στην Κίνα βρίσκονται. Ή μήπως ε, στην κατανάλωση στα καταστήματα. Πού βρίσκονται αυτά. Λοιπόν, δεν είναι απλό να καθοριστεί. Αυτό που ξέρω είναι το εξή. Αν δεν τα πάμε καλά τώρα, αν δεν το πετύχουμε τώρα, θα βλάψουμε την δυνατότητα της Ευρώπης να μπει στην ψηφιακή οικονομία και θα βλάψουμε κυρίως τις οικονομίες και τις χώρες που είναι πρώτες και καλύτερες στην ψηφιακή οικονομία. Εκτιμώ τη δουλειά των εισηγητών και των συνεισηγητών, αλλά πιστεύω ότι από πλευρά μου τουλάχιστον τα έχουν περιπλέξει παραπάνω τα πράγματα και αυτό επειδή είναι περίπλοκη η πραγματικότητα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα αυτό. Αλλά είναι δύσκολο να οριστεί ως ευέλτιστη η τρέχουσα κατάσταση είναι κάτι λιγότερο αποβέλτιστη. Πώς να το κάνουμε σε ό,τι αφορά και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού κτλ. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση με ένα εργαλείο ανταγωνισμού κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός, ο δίκαιος ανταγωνισμός. Και θεωρώ ότι και αυτός είναι ένας τρόπος ε, να το κοιτάξουμε το θέμα. Ο κύριος Σαΐς είναι ο Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και να συμφωνήσω με τους συναδέλφους και να συγχαρώ τους εισηγητές, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Και υποπτεύομαι ότι η συζήτηση στην Επιτροπή μας και η ποικιλία, η διαφορά, αν θέλετε, των ε, απόψεων που εκφράζονται αποτυπώνουν και τον κοινωνικό ιστό γιατί όλοι θέλουν προφανώς και μικρέ και μεγάλες επιχειρήσεις να πληρώνουν τα όσα τους αναλογούν σε φόρους. Όλοι θέλουμε φορολογική διαφάνεια, όλοι θέλουμε να καταπολεμήσουμε τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Αυτό αποτελεί τμήμα δημοκρατικής κοινωνίας. Όλοι αυτό θέλουμε να το πετύχουμε. Άρα το πώ θα το πετύχουμε, αυτό είναι που συζητάμε ε, σήμερα. Εγώ πιστεύω περιπαθώς, Πρόεδρε, ότι οι επενδύσεις στην Ευρώπη, οι άμεσες επενδύσεις ε, στην Ευρώπη από άλλα μέρη του κόσμου, συνδέονται άρρηκτα με την φορολογική συνοχή και συνεκτικότητα και μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις θα θέλουν να επενδύουν στην Ευρώπη αν υπάρχει ένας συνεκτικός και διαφανής φορολογικός συντελεστής και φορολογικό σύστημα. Δηλαδή, ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα. Και όπως λοιπόν διαπιστώνουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διάφορα κρατημέλη έχουν διαφορετικές πολιτικές και αυτό αποτελεί προφανώς απορία της δικής τους ιστορία, της δικής τους οικονομικής πολιτικής. Εγώ είμαι από μια χώρα που μέχρι την δεκαετία του 60 ήταν μια οικονομία ουσιαστικά γεωργική, αλλά ουσιαστικά επέλεξε. Επέλεξε να χρησιμοποιήσει την ανάπτυξη FTI και μια μεγάλη, τεράστια, ένα τεράστιο δυναμικό εξαγωγών για να α, επαναπροσδιορίσουμε την οικονομία μας. Αυτή την οδό α, ακολουθήσαμε και όταν ήμουν στην κυβέρνηση στην Ιρλανδία υπήρξε μεγάλη πίεση, τεράστια πίεση να αλλάξουμε τον εταιρικό φορολογικό κώδικα τότε και είχαμε πει τότε ότι ο καλύτερο τρόπο να μείνουν οι επενδύσει στην Ιρλανδία και στην Ευρώπη είναι να εξασφαλίσουμε ότι είναι ξεκάθαρο, συνεκτικό και ενιαίο το θέμα του φορολογικού συντελεστή. Αυτό και έγινε. Και ο λόγο για τον οποίο έχουν ουσιαστικά διπλασιαστεί οι φορολογικοί συντελεστέ στην ε, Ιρλανδία τα τελευταία 6 χρόνια δεν έχει να κάνει με την ανα αν θέλετε, με την ε, να διαπραγματεύσει τη οικονομία έχει να κάνει και με τα PEPs του ΩΣΑ. Λειτουργούν. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα παίρνουμε πιο πολλά φορολογικά έσοδα από τι μεγάλε εταιρείε, γιατί ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός αντιμετωπίζεται σε επίπεδο ΩΣΑ σήμερα και αυτή είναι η καλύτερη οδό αν πραγματικά θέλουμε να επιλύσουμε το θέμα αυτό. Πιστεύω Πιστεύω, όπως ο κ. Χόκμαρκ, ότι η φορολογική πολιτική αποτελεί λειτουργία των επικυρίαρχων δημοκρατικών κρατών. Ο φορολογικό ανταγωνισμό πιστεύω ότι είναι καλό πράγμα και πιστεύω ότι το να μείνουν οι επενδύσεις και τα ταμεία στην Ευρώπη, ο ανταγωνισμό με ε, τις άλλες χώρες δεν είναι μια ισοπαίδωση των όρων είναι υγιής ανταγωνισμός. Πώς θα προσελκύσουμε εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα το συζητήσουμε προφανώς, θα το έχουμε υπόψη, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι απόλυτα θετικό, ιδιαίτερα για τα μικρά κράτη-μέλη, τα οποία δεν έχουν μια τεράστια βιομηχανική παράδοση που πρέπει να δώσουν ένα καινούργιο νόημα και μια νέα κατεύθυνση στην οικονομία τους, σε αντίθεση με τις μεγάλες χώρες, τις τεράστιες χώρες που έχουν τεράστια εσωτερική κατανάλωση, μιας και η οικονομία του λειτουργεί έτσι. Αυτό δεν ισχύει σε μικρές ε, χώρες όπου εξορισμού έχουν πιο πολλές εξαγωγές και άρα προσαρμόζονται πιο πολύ Στι οικονομικές εξελίξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι ο φορολογικό ανταγωνισμό είναι φωτικό. Δεν έχω εγώ τέτοια ιδεολογικά ζητήματα. Πιστεύω ότι είναι ο καλύτερο τρόπο να παραμείνει σε επαγρύπνηση η Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα πρότυπα αυτά. Ένα άλλο σχόλιο καταλεκτικό. Αυτή η συζήτηση λοιπόν την ξεκινάμε χωρίς καμία συνεννόηση για τις ενδυνάμει αρνητικές συνέπειες που θα υπάρξουν για τη φορολογική βάση κάθε κράτο μέλου. Αυτό δεν βλέπω δεν, δεν μου φαίνεται σωστό. Παρά αυτά που ακούμε για μια επιτροπή αποζημίωση και τα λοιπά, όλα αυτά τι να σας πω, μου ακούγονται λίγο σοσιαλιστικά, δεκαετία του 50 ότι μπορούμε δηλαδή να δώσουμε αποζημίωση για τις ζημίες και τα λοιπά. Στη χώρα μου αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την φορολογική βάση μέχρι και ένα τρίτο. Εγώ αυτό που θέλω να ξέρω λοιπόν και θέλω να ξέρω και οι εκλογέ μου, ποιος θα τα πληρώσει, ποιος θα πληρώσει τη διαφορά αυτή. Αν υπάρχει διαφορά δηλαδή στη φορολογική βάση στην Ιρλανδία 2 δισεκατομμυρίων, ποιο θα τα πληρώσει όλα αυτά για τα μεγάλα κράτη-μέλη που έχουν τεράστια ιστορική οικονομία και μπορούν να παίξουν ε, με τέτοια πόσα. Ε, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα αλλά για τις μικρές, εταιρείες, ε, τις μικρές χώρες αυτό σημαίνει τεράστιες διαφορές. Προσπαθήσαμε λοιπόν στις τροπολογίες μας να τα αποτυπώσουμε αυτά, να σας ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τον κύριο Φέρπερ και τους άλλους που εξετάζουν τις τροπολογίες, αλλά να έχουμε ένα ρεαλισμό στην ουσία για την ε, τοποθέτηση των οικονομιών μας με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Γιατί τότε πιστεύω ότι θα πετύχουμε πραγματικά ένα αποτέλεσμα δίκαιο για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο στη συζήτηση, αλλά ακούγοντα τον συνάδελφό μου που τον προκαλήσαντα, ε, αισθάνθηκα ότι πρέπει να μιλήσω. Ε, δεν είμαι γνωστή ω κάποια που είναι υπερθερμα... που υπερθεματίζει υπέρ του παλιού σοβιετικού μοντέλου ούτε ε, είμαι θειασότης επίσης ε, του άκρατου ας πούμε ανταγωνισμού ως το α και το ω της οικονομικής πολιτικής. Αλλά σε αυτή τη συζήτηση θέλω να τιμήσω αυτή τη βασική αρχή της ε, συνθήκης ε, της Ρώμης ε, που υποστηρίζουν και διάφοροι συνάδελφοι του ΕΛΚΑ. Δηλαδή της αρχής του απρόσκοπτου και μη στρεβλωτικού ανταγωνισμού. Με σοκάρει το γεγονός που ακούω διάφορα σήμερα. Δεν ξέρω καν πότε δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα εργασία κυρία Πριμαρόλο πριν ακόμα τον κώδικα διοντολογίας ούτω ώστε να μιλήσουμε για αυτόν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το μη στραβλωτικό μεταξύ των κρατών μελών. Και πώ να μην αναγνωρίζουμε ότι μέσω αυτή τη αρχή, την οποία αγνοούμε εντελώ. Έτσι. Πώς εξηγείται ότι τελικά καταλήξαμε να, να ανακαλύπτουμε, μάλλον αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε χθε και προχθές πούμε, όλα αυτά τα εξωφρενικά που μας ε, παρουσίασαν διάφοροι πολύ ε, θαραλέοι δημοσιογράφοι. Το πρώτο μάθημα από, τα Panama Papers, που επιβεβαιώνεται από τα Paradise Papers, είναι ότι χρειαζόμαστε το CCCTB. Ακούμε να μας λένε ότι τα μεγάλα κρατημέλη δεν έχουν μια στρατηγική ανάπτυξη ε, ανάπτυξης που ε, να, συνδέεται με την εσωτερική τους αγορά. Εγώ ξέρω μια μεγάλη ε, τέτοια χώρα που είναι στραμμένη προς τις ε, ε, εξαγωγές ε, που έχει καλή όμως φορολογία με σωστή φορολογική βάση κτλ. Πρέπει να απαντήσουμε στο εξή ερώτημα. Εάν όλα είναι καλά, τότε γιατί φτιάξαμε φορολογικούς συντελεστές τους πιο χαμηλούς δυνατούς. Και ξέρετε ότι ακριβώς αυτού του τύπου οι φορολογικοί συντελεστές οδήγησαν σε αυτά τα Panama Papers. Ε, και μία από αυτές τις εταιρείες που επωφελείται από αυτούς τους συντελεστές είναι η, Apple. Εγώ ανησυχώ λιγάκι. Φυσικά τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν αυτά που, κάνουν ε, στο παρελθόν, ε, που δεν θέλουν να αλλάξουν, υπάρχουν αντιστάσεις, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Άκουσα το, από την άλλη όμως ε, αυτό που είπε ο κ. Χόκμαρ ότι κάποιες χώρες θέλουν να πληρώσουν περισσότερα για τις δημόσιες υπηρεσίες ε, και είναι δική τους επιλογή. Ε, και σε αυτή την περίπτωση α προσελκύσουν ξένα κεφάλαια. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί χρειαζόμαστε τα ξένα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τι δημόσιε επιχειρήσει, γιατί ακριβώ χαμηλώνουμε τόσο πολύ του φορολογικού συντελεστέ, μειώνει τόσο πολύ τα φορολογικά κέρδη που χρειαζόμαστε αυτά. Ε, εγώ πιστεύω ότι αυτέ οι δύο πολύ καλέ εκθέσει θα μα επιτρέψουν να προχωρήσουμε να έχουμε μια επιθετική στάση απέναντι στο Συμβούλιο και θα μας επιτρέψουν ακριβώς να απαντήσουμε σε αυτά τα προβλήματα. Να στραφούμε και να μπορούμε να σταθούμε προς αυτούς εκλογικούς μας και να πούμε ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα ας πούμε, δεν τα αντιμετωπίσαμε σαν να είναι τίποτα. Δεν μπορείτε να πείτε ότι αυτή η θαυμάσια δουλειά που κάνουν οι δημοσιογράφοι, όλα αυτά τα σκάνδαλα που αποκαλύπτουν, α πούμε, εμά μα αφήνουν να τους και ότι δεν αλλάζει καθόλου η δουλειά μα. Δεν επηρεάζουν καθόλου τη δουλειά μα. Ε, είναι μια ευκαιρία αυτή που μα δίνεται για να συμφιλιώσουμε να συμφιλιώσουμε τα κράτη-μέλη, να υπάρξει ένας δίκαιος, μια δίκαιη έτσι φορολόγηση στα κράτη-μέλη, ε, συνέπεια και διαφάνεια. Και η διαφάνεια και συνέπεια τι σημαίνει. Να έχουμε μια κοινή ενοποιημένη βάση. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της οικονομίας. Δηλαδή ενσωματώνοντας ε, την ιδέα της μόνιμης εγκατάστασης ε, που φυσικά δεν υπήρχε αυτή η έννοια ε, όταν... όταν δημιουργήσαμε τα φορολογικά καθεστώτα που ξέρουμε σήμερα. Uh, Ευχαριστώ. Ο Διευθυντή στην Γενική Διεύθυνση Ταξούντα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Ε, Κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, χαίρομαι που θα πω και εγώ δύο λόγια για αυτή τη συζήτηση για το CCTB και CCCTB. Όχι για να ανακατευτώ στις δικές σας εργασίες, αλλά για να σας πω την εκτίμηση, την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η οποία θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο κάνει πολύ καλή δουλειά. Το αποδεικνύει και η σημερινή συζήτηση. Καταρχάς, Είμαστε υπέρ της προσέγγισης των εισηγητών. Να αντιμετωπίσουμε τα δύο θέματα από κοινού. Παράλληλα, η ιδέα του να χωρίσουμε την πρόταση του 2011 δεν ήταν ε, δική μας επιλογή, ε, δεν το κάναμε γιατί το θέλαμε, ήταν, έγινε για λόγους έτσι λογικής ας πούμε. Γιατί ακούσαμε τα επιχειρήματα που, υπήρχαν στο Συμβούλιο, ήταν δύσκολο να διαπραγματευτούμε ε, με τη μια και τα δύο αυτά σχέδια. Ε, δεν μπορούσε το Συμβούλιο. Το θεωρούσε δύσκολο. Επίσης, συμφωνούμε με την προσέγγιση κατά την άποψη ότι τα ωφέλη από τις ε, δύο προτάσεις προκύπτουν κυρίως από τη φάση της ενοποίησης, η οποία θα πρέπει να προκύψει πολύ πολύ γρήγορα μετά τον καθορισμό της βάσης, τη φορολογικής βάσης. Πρώτα φορολογική βάση ποια είναι, ας πούμε, και μετά ενοποίηση. Επίσης, το στοιχείο της ενοποίησης είναι το στοιχείο το οποίο φέρνει τα περισσότερα ωφέλη στους δύο στόχους που θέλουμε να υλοποιήσουμε με τις προτάσεις. Δηλαδή, ε, μείωση της φορολογικής βελτιστοποίησης, αλλά να υπάρξει και ένα καλό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις ε, με την ενοποίηση σε ό,τι αφορά την μείωση του κόστους ε, που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις λόγω του ότι έχουν ε, να αντιμετωπίσουν 28 διαφορετικά φορολογικά συστήματα επιτυγχάνεται. Επίσης, αυτό ήταν ένα σημαντικό θέμα. Είναι σημαντικό επίσης και οι διάφορες τροπολογίες μπορούν να εξυπηρετήσουν πάρα πολύ αυτό το στόχο. Εμείς πολύ γρήγορα αναγνωρίσαμε ότι μπορεί να βελτιωθεί φυσικά η πρόταση της Κομισιόν Ήμασταν πολύ ανοιχτοί από την αρχή να εξετάσουμε αυτές τις βελτιώσεις. Επ' θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πολ Τάν και τον Αλέν Λαμασού για τη δουλειά που κάνανε, για την προσωπική τους έτσι, ανάμιξη, για τη διαθεσιμότητά τους να συμμετάσχουν στις διάφορες διασκέψεις και συναντήσεις. Επίσης, ε, του ευχαριστώ και για την ασθενή σχέση που είχαμε τα διάφορα ε, εθνικά κοινοβούλια. Είναι ένας φάκελος που παρουσίασε η Κομισιόν με σεβασμό τη αρχή της αναλογικότητας και επικουρικότητα και που βρίσκεται στην καρδιά βεβαίω της οικονομικής και φορολογικής πολιτικής των κρατών μελών. Και το να έχουμε μια έντονη σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια για να τους εξηγήσουμε την προσέγγιση μας, αλλά για να ακούσουμε τις απόψεις τους και τις δυσκολίες που έχουν, τόσο ώστε να τις λάβουμε υπόψη και να βρούμε λύσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Στα πλαίσια των εργασιών σας υπάρχουν διάφορα στοιχεία βελτιωτικά που προτείνονται και που κατά την άποψή μας πραγματικά κινούνται προς την κατεύθυνση. Καταρχάς, το σύνολο του πακέτου που αφορά με την ε, ψηφιακή οικονομία ή την ψηφιοποίηση της οικονομίας μας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και η Κομισιόν ε, αποφάθηκε από αυτού στις 20 Σεπτεμβρίου μέσω μιας ανακοίνωσης και είμαστε σε φάση που το δουλεύουμε ακόμα. το δεν είναι, γνωστό σε όλους ότι το διαφθορτικό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, της φορολόγησης των επιχειρήσεων ε, με την ψηφιοποίηση της οικονομίας είναι ακριβώς το CCCTB. Γι' αυτό οποιαδήποτε βελτίωση, είτε στον ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης, είτε στη βελτίωση του price ε, transfer, transferring, δηλαδή της μεταβιβαστικής τιμολόγησης. Όλα αυτά ε, οι τύποι για την κατανομή της ενοποιημένης φορολογικής βάσης, όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Επίσης, διάφορες συζητήσεις για τα κατόφλια το πώ αντιμετωπίζουμε τι διάφορε απομειώσει και εκπτώσεις των διαφορών ταπανών ή βαρών ας πούμε, που έχουν οι επιχειρήσει. Παραδείγματο χάρη για την έρευνα και την κοινοτομία. Ή η μεταφορά από χρόνο σε χρόνο των ζημιών, ας πούμε. Όλα αυτά τα στοιχεία ε, θα πρέπει να τα συζητήσουμε και να, φυσικά θα πρέπει καταρχάς να συμφωνήσουν διάφορες πολιτικές ομάδες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλούς ορισμούς για την ε, φορολογική βάση, η φορολογητέα βάση. Τελευταίο σημείο τη παρέμβασή μου. Αυτό που έχει σημασία είναι τι θα ισχύσει από τώρα, από εδώ και πέρα. Καταρχάς, να δούμε μαζί τα δύο θέματα, τους δύο φακέλους. Όπως είπαν και διάφοροι συνάδελφοι, καλό είναι να το αντιληφθεί το Συμβούλιο ως μια πολύ λογική βάση για να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις για τα δύο θέματα μαζί. Επίση, Επίσης, ε, βραχυπρόθεσμα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει στην, στο Συμβούλιο και το θέλει η Εστονική και η επερχόμενη Βουλγαρική Προεδρία να υπάρξει μια σταθεροποίηση της φορολογικής βάσης, φορολογητέας βάσης. Γιατί είναι το αρχικό σημείο στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε για να γίνει καλή συζήτηση με τα κράτη-μέλη. Για να δούμε τι επιπτώσει θα έχει αυτή η εναρμονισμένη βάση στα φορολογικά του έσοδα. Ε, αυτό το κάνουμε μαζί με τα κράτη-μέλη. Είναι μια πολύ σημαντική συνεργασία. Γιατί μόνο έτσι θα, δούμε, ε, θα κάνουμε μια καλή αποτίμηση ας πούμε, των επιπτώσεων στα φορολογικά έσοδα. Και επίσης, αν ο τύπος ε, για την ε, ενωπημένη φορολογική βάση θα πρέπει να επανεξεταστεί. Πολύ σημαντικό αυτό. Τέλος, το θέμα των συντελεστών. Πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η θέση της Κομισιόν ήταν πάρα πολύ σαφής από την αρχή, από την ανακοίνωση που βγάλαμε το 2015 για το θέμα αυτό. Ε, υπερασπιζόμαστε την αρχή μιας ενός φορολογικού ανταγωνισμού υγιούς και διαφανούς στην ε, εσωτερική αγορά. Ακριβώς γι' αυτό πιέζουμε για να υπάρχει ακόμα περισσότερη διαφάνεια. Ακριβώς γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν προτείναμε μία εναρμόνιση των συντελεστών, των φορολογικών συντελεστών δηλαδή, για τον εταιρικό φόρο. Θέλουμε να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός επί, της επί τη βάση μιας ε, Εναρμονισμένη ε, φορολογική βάση, ενώ του φορολογικού συντελεστέ θα του καθορίζουν ε, ελεύθερα τα κράτη-μέλη. Ε, επίσης, μα γι' αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε ε, υγιή ανταγωνισμό και θα έχουμε και καλές φορολογικές συμφωνίες. Αυτά και περιμένω με ανυπομονωσία την ε, ολοκλήρωση των εργασιών σας. Είναι η απαρχή της συνέχισης της συνεργασίας μας και συνεχεία βεβαίως μετά τις δικές εργασίες θα ξεκινήσει και η μεγάλη συζήτηση στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα οι εισηγητές παρακαλώ έχουν το λόγο. Ο κύριος Λαμασούρ. Πρώτος. Δεν ξέρω τι προτιμάτε. Ο κύριος Τάγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω να πω ότι δεν είμαι από μικρή χώρα. Να διευκρινίσω αυτή την παρανόηση. Είναι τεράστια η Ολλανδία στη φοροαποφυγή. Για παράδειγμα, Λουξεμβούργο και Ολλανδία η φοροδιαφυγή είναι τεράστια. Στην Ιρλανδία λοιπόν, να σας πω, έχουμε πιο πολλές μεγάλες άμεσες επενδύσεις από ότι η... Γαλλία και η Γερμανία. Ξέρετε τι είναι αυτό όμως. Αυτό είναι φορολογικός σχεδιασμός, είναι χαρτιά. Δεν έχει να κάνει αυτό με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Και η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο έχουν μεγαλύτερες άμεσες επενδύσεις ε, σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Αυτά είναι χαρτιά όμω. Σα λέω λοιπόν, επειδή θέλετε διαφάνεια, ποια είναι τα διαφάνεια ποια είναι η διαφάνεια, ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία. Και αυτό καταδεικνύει τι κάνουν οι μικρές χώρες. Καταχωρίζουν ε, τις άλλες χώρες ε, ως φορολογική βάση. Πειρατεία, πειρατεία είναι αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει καταργηθεί πριν από δεκαετίες πριν από αιώνε. Και γι' αυτό λοιπόν τίθεται το θέμα τη επικορικότητα. Γιατί αν μείνουν τα πράγματα έτσι, δεν θα σταματήσει η πειρατεία. Πού λοιπόν τίθεται το θέμα επικυριαρχία, αν δεν υπάρχει καμία χώρα που να επιλέγει υψηλότερου ευρωλογικούς συντελεστέ. και όλοι επιλέγουν χαμηλότερους. Πού λοιπόν θα γίνει η συζήτηση. Περιμένω λοιπόν πραγματικά από τις μεγάλες χώρες να μπουν πρόδρομοι και να σταματήσουν αυτή την πειρατεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μοναδικός τρόπος που θα λειτουργήσει η κατάσταση αυτή γιατί η δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Δεν θα σταματήσουν οι κάτω χώρες. Και θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση στην τρέχουσα κατάσταση γιατί όπως είπε ο πρόεδρος δεν είναι σε καμία περίπτωση ιδανική η κατάσταση. Όλα αυτά τα κρατημέλη που πλήττονται δεν ήταν σε θέση να ε, μπουν σε ψηφιακές πλατφόρμες, Facebook, Google, τη γλιτώνουν και δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους. Έχουμε χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο φορολογούμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει πέντε σύμφωνα με τις αξιολόγησεις μας και τις εκτιμήσεις μας λόγω της πειρατείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μη μας λέτε να τα κάνουμε αυτά στον ΩΣΑ. ευχαριστώ να έβρισκε ο ΩΣΑ μια διεθνή λύση. Αλλά το πρώτο σημείο δράση στην ΠΕΠΣ δεν είναι δράση, είναι αδράνεια, έλλειψη δράσης, παράταση για πέντε χρόνια. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την φορολογία της ψηφιακής εικόνα μας. Άρα όσα την Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει να ηγηθεί αλλιώς, δεν θα, ξανα... δεν θα βγούμε από την κατάσταση αυτή ποτέ από το φαύλο κύκλο. Θα πρέπει να φορολογηθεί και η Google και η Facebook. Και πώς θα γίνει αυτό αν δεν είναι ευρωπαϊκές. Δεύτερο θέμα, ο φορολογικός ανταγωνισμός που βλέπουμε τώρα είναι προς όφελος των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων ομίλων και ε, δεν ευνοεί τις μικρόμεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι σωστό λοιπόν και δεν οδηγεί σε δίκαιους όρους ανταγωνισμούς. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αναλογικά 30% μεγαλύτερο φιλογικό φορτίο σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες. Δεν είναι σε καμία περίπτωση δίκαιο αυτό και σίγουρα δεν θέλουμε τέτοιο ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό λοιπόν είμαστε σαφείς και από αυτού. Και χαίρομαι, χαίρομαι ιδιαίτερος που προτείνεται από διάφορους συναδέλφους να φορολογηθεί η ψηφιακή οικονομία, γιατί πιστεύω ότι αποτελεί πολύ πιστικό πρόβλημα. Και θα ήθελα να πω με πάσα σαφήνεια ότι δεν πιστεύω ότι ο φόρος επί του κύκλου εργασίων. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να βρείτε μία λύση βέβαια, αλλά πιστεύω ότι πρόκειται για μία αδρή και ad hoc λύση σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο. Γιατί να μην ξεκινήσουμε με μια ενιαία κοινή αναπημένη βάση φορολογικής προλόγησης. Ε, Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να φορολογήσουμε την Apple, την Google, την Facebook. Και συμφωνώ τέλος ότι αν θέλουμε τέτοια λύση και βλέπουμε ότι κάποιες χώρες μπλοκάρουν ακόμα τέτοιες λύσεις. Θα πρέπει να κοιτάξουμε σίγουρα τη λύση της ενισχυμένης συνεργασίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα αφήσουμε έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει κάποιες χώρες να μπουν πρώτες και να δείξουν ότι μπορεί να αλλάξει ο κόσμος της φορολογίας και ότι μπορούν να δοθούν πρότυπα για να αλλάξει πραγματικά η φορολογική κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κ. Λαμασού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τις ε, απόψεις τους, τις επικρίσεις, τις τροπολογίες ε, που εμπλουτίζουν τη συζήτηση. Και πράγματι η συζήτηση αυτή ήταν ε, εξαιρετικού επίπεδου πάνω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μετά τις ε, παρατηρήσεις του Πολ που τις εξέφρασε με πολύ δυναμικό τρόπο, συμφωνώ απόλυτα μαζί του, θα ήθελε να ε, επιμείνω σε τρία ζητήματα. Πολύ ωραία ξεκινάει ο Νοέμβριος. Ο Μάρκους Φέρμπερ ήταν ο πρώτος που σύστησε να διατηρήσουμε στενή συνεργασία, στενή επαφή με τον ΩΣΑ, κυρίως αν θέλαμε να ξεκινήσουμε καινοτομίες όπως ε, η, τα μέτρα σχετικά με την ψηφιακή οικονομία. Όπως είπε όμως και ο Πολ, ο, ο ΣΑ προχωρεί πολύ προσεκτικά και δεν θα λάβει καμία πρωτοβουλία. Αν όμως εμείς λάβουμε πρωτοβουλία πρωτοβουλία ρεαλιστική φυσικά και ε, λογική που ε, αντιστοιχεί στην ε, σημερινή ψηφιακή οικονομία. Τότε θα αποτελέσει μια τέτοια πρωτοβουλία σημείο αναφορά για τον όσα. Να υπενθυμίσω ότι υπό τη γερμανική προεδρία του G20 το G20 ζήτησε από τον ΩΣΑ να κάνει προτάσεις σχετικά με την φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρήσεων και φυσικά το ίδιο έκανα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, απευθύνθηκε στο, ε, στην Κομισιόν. Την ερχόμενη άνοιξη λοιπόν θα καταβληθούν προτάσεις και αν μέχρι τότε το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει καταθέσει αν μέχρι τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταθέσει μια λογική πρόταση, θα συμβάλλει σημαντικά στην πολιτική συζήτηση και στις εξελίξεις. Το δεύτερο, ο ελάχιστος συντελεστής. Ε, ε, είναι σαφές ότι Παραδοσιακά αντιτίθενται η αριστερά και η δεξιά σε ένα τέτοιο θέμα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το Συμβούλιο δεν θα δεχτεί ποτέ μια εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών. Κάτι τέτοιο πάει πολύ μακριά σε ό,τι αφορά την ε, κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στη κράτη-μέλη και την Κομισιόν. Η φορολογία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλό να εναρμονίσουμε τον ορισμό του φορολογητέου κέρδους. Δεν πιστεύω όμως προσωπικά ότι μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή. Ο ελάχιστος συντελεστής για πολιτικούς λόγους, για παράδειγμα 18-20%, ε, επειδή είναι πολιτική επιλογή. Δεν είναι δική μου επιλογή, ούτε ε, της ομάδας μου, αλλά καταλαβαίνω ότι τέτοια επιλογή κάνουν άλλοι συνάδελφοι, άλλες ομάδες. Υπάρχει και ο ελάχιστο συντελεστή από τεχνική απόψεω. Γιατί αν πούμε ότι δεν υπάρχει ελάχιστο συντελεστή και κάποιο κράτο μέλο ε, επιλέξει 1,5% φορολόγηση, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου φορολόγηση. Μπορούμε, πιστεύω, να βρούμε ένα συμβιβασμό σε ό,τι αφορά τον ελάχιστο συντελεστή από τεχνική απόψεω. Θα ήθελα όμω να επιστήσω την προσοχή ε, σε ακριβώ αυτή τη διάθεση. Και μία τελευταία παρατήρηση ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση ε, με πρωτοβολία διαφόρων συναδέλφων και φίλους από τον ΕΛΚ. Σε ό,τι αφορά το αν είναι θεμητό ή όχι να παρέμβουμε σε νοσιακό επίπεδο προκειμένου να ε, εναρμονίσουμε, να καταλήξουμε στην εναρμόνιση του ορισμού του φορολογητέου κέρδους. Κάθε φορά ότι, ε, που ακούω για μικρό κράτος μέλους, υποψιάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι κάποιες χώρες μπορούν να πληγούν και κάποιες άλλες όχι μια μικρή χώρα που μπορεί να υποφεληθεί από μια μικρή ε, αγορά και πρέπει να βρει τρόπο να ευημερήσει και με άλλους τρόπους, αυτά ακούγονται. Μια μικρή χώρα όμως έχει πρόσβαση στην ίδια αγορά με όλες τις χώρες, με 500 εκατομμύρια κατοίκους, πολίτες. Χάρη στην ενιαία αγορά όλα τα κράτη-μέλη εποφελούνται από την ίδια ε, αγορά τις ίδιες υπηρεσίες. Μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε παορίστου για τις, ε, τα πλεονεκτήματα των μικρών και των μεγάλων κρατών μελών. Είμαστε περήφανοι που έχουμε μεγάλα κράτη-μέλη, μικρά κράτη-μέλη και λεγόμενα μεγάλα κράτη-μέλη, γιατί έχουν περισσότερους πολίτες. Όπως είπε ο Ζων Κλοντ Κλοντ-Γιούγκερ, υπάρχουν δύο ε, είδη κρατών μελών, δύο κατηγορίες, αυτοί που ξέρουν ότι, αυτά που ξέρουν ότι είναι μικρά και αυτοί που θεωρούν ότι είναι μεγάλα. Ανάλογα με το σύστημα που εφαρμοστεί, ίσως κάποια κράτη χάσουν φορολογικά έσοδα και θα πρέπει να βρούμε τρόπους αντιστάθμισης και έχουν κατατεθεί οι και φυσικά είμαστε ανοιχτοί στι δυνατότητε βελτίωση τη πρόταση που έχουμε καταθέσει. Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση της ψηφιακή οικονομίας, θα ήθελα ε, να σας να καθισχάσω το, συνάδελφο λέγοντας ε, το εξής. Πήγαμε με το Πολ στο ε, Ταλίν και όταν συναντήσαμε τον αρμόδιο υφυπουργό στις αρχές του καλοκαιριού μας είπε πολύ φιλικά το CCTB ε, δεν ε, συμφωνούμε ιδιαίτερα στην Εσθονία. Έτσι λοιπόν παίξαμε το παιχνίδι και φυσικά εντάξαμε το θέμα στην πολιτική ατζέντα προκειμένου να βρεθεί ε, μια συμβαστική λύση μέχρι το τέλος της εθνικής Προεδρίας. Πάντως επιμένουμε να ενταχθεί στο CCTB η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Η Εσθονία βασίζεται στην ψηφιακή οικονομία και είναι ξεκάθαρο σαφές ότι αν οι Εσθονοί μας είχαν πει κάτι τέτοιο δεν γίνεται με τίποτα, ίσως να είχαμε διαφορετική ε, συμπεριφορά. Μας ενθαρρύνουν οι Εσθονοί. Και σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, προλαλήσαντες είπαν ότι στη σημερινή ψηφιακή οικονομία ξέρω ξέροντας ότι δεν, θα, δεν γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον από την άποψη των ψηφιακών εξελίξεων. Μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Όλες οι διαβολεύσεις που έγιναν, όλα όσα διαβάσαμε δείχνουν ένα πράγμα. Υπάρχει ένα μόνο πράγμα που δεν μπορεί να μεταγκατασταθεί. Τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά μου προσωπικά δεδομένα που δίνω δωρεάν στο, στη Facebook. Facebook μπορεί να τα συλλέξει και να τα επεξεργαστεί ε, οπουδήποτε στον κόσμο, ακόμα και σε ένα ε, υπολογιστικό νέφος. Γι' αυτό κάναμε αυτές τις ε, προτάσεις. Και κάτι τελευταίο, το θέμα της επικουρικότητας και ε, το ότι η φορολογία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πρέπει να, ξεκα... ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην επικουρικότητα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Ναι, η αρμοδιότητα, η φορολογία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και είμαι έτοιμος να το υπενθυμίσω στην έκθεση αν ε, υπάρχει τέτοια βούληση. Είναι το πρώτο πράγμα που ε, τονίζουμε κάθε φορά που συναντούμε εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σε κάθε συνέντευξη τύπου. Και αυτό ακριβώς θα ξαναπούμε μεθαύριο στη Σόφια. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο της ενιαίας αγοράς είναι αρμοδιότητα της Ένωσης και προβλέπει η συνθήκη άρθρα που ε, συνδυάζουν τα δύο θέματα. Πρέπει να το συζητήσουμε φυσικά. Δεν μπορεί μια αγορά, μια ενιαία αγορά να λειτουργήσει με εναρμενισμένο τρόπο, με μια, ένα ενιαίο νόμισμα και μια ενιαία πολιτική σε διάφορα θέματα, αλλά ε, δεν έχει επαρκή εναρμόνιση σε ό,τι αφορά τον τομέα της φορολόγησης των εταιριών. Υπάρχει και απ' την άλλη το θέμα της επικουρικότητας. Η επικουρικότητα δεν σημαίνει ότι εξετάζουμε τα ε, προβλήματα στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Η επικουρικότητα σημαίνει ότι εξετάζουμε τα προβλήματα στο κατάλληλο επίπεδο και όταν καλούμαστε να διαπραγματευτούμε με μια πολυεθνική που μπορεί να έχει ένα τζίρο, μια κεφαλοποίηση ή κέρδη ε, που υπερβαίνουν ε, το ΕΠ ενό κράτους μέλους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τριπλάσια του ΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας είναι καλύτερα οι διαπραγματεύσεις να γίνουν σε ενωσιακό επίπεδο και όχι σε εθνικό επίπεδο. Ας μην ε, τερματίσουμε τη συζήτηση σήμερα. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία. Θέλουμε να καταθέσουμε μία πρόταση που θα οθήσει το Συμβούλιο Υπουργών να προχωρήσουν προς μία συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ του συζήτητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και του υπόλοιπου μιλητέ και νομίζω ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη και σημαντική η συζήτησή μας. Εγώ προσωπικά συμφωνώ ιδιαίτερως με τα συμπεράσματα και των δύο εισηγητών ε, και φυσικά θα αποφανθεί και η Επιτροπή σύμφωνα με τη συνήθεια διαδικασία. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2018 θα μεταβούμε στην Ολομέλεια. Αυτό είναι το σχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. We are five minutes earlier, four minutes earlier. Έχουμε και τέσσερα λεπτά χρόνο, λέει ο Πρόεδρος. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε, φαντάζομαι. Εδώ είναι και ο κύριος Τόλογιαν. So, uh, maybe we will make then a suspension in case... Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. If needed, let's see. And, uh, let's prepare papers. Sorry, I invaded you.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 So, Μάλιστα και περνάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, ε, εξέταση του σχεδίου έκθεσης ε, για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματο σε τιμές αγοράς. Κανονισμός ΑΕΕ. Εισηγητής ο υποφανόμενος. Εξ ονόματος λοιπόν του Προεδρείου. σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης, το οποίο και έχω προετοιμάσει. Το νέο νομικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της Λισαβόνας και την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε πιο διαρθρωμένες και στοχευμένες προσεγγίσεις, ούτως ώστε να έχουμε δεδομένα για το ΑΕ πιο αξιόπιστα, ε, απέτησαν την αναθεώρηση του προηγούμενου κανονισμού του Συμβουλίου του 2003. Η αξιολόγησή μου για την πρόταση της Κομισιόν είναι γενικά θετική. Έχει σαν σκοπό να ενισχύσει την συγκρισιμότητα, αξιοπιστία και πληρότητα των συνολικών στοιχείων ΑΕ πάνω στο οποίο βασίζεται βασίζονται οι διπόροι μας. Επίσης, το άρθρο 338 τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η νέα νομική βάση, είναι απόλυτα λογική, απόλυτα ενδεδειγμένη, όχι μόνο λόγω της αλλαγής που προέκυψε στην απόφαση για τους ιδίους πόρους, αλλά και γιατί τα δεδομένα για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα ε, χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέρα από τους ίδιους πόρους και για να υπάρξει στατιστική ακαιρεότητα και πληρότητα. Ο στόχος της πρότασης συνάδει με τους στόχους της ανακοίνωσης του 2011 για τη μεθοδολογία για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών ε, της επόμενης δεκαετίας που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και την, ε, και την ε, στατιστική, στατιστικά δεδομένων μέσω ε, δεδομένων για τους ίδιους πόρους. Η προσαρμογή στους ορισμούς ε, στα νέα λογιστικά πρότυπα για το, τους ίδιους πόρους, ε, ουσιαστικά για το ΑΕ και για τη συγκρισιμότητά του, θα βελτιώσει και την πολιτική που χρησιμοποιούμε, αλλά θα δώσει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν το παλιό σύστημα του 1995 καθώς και το σύστημα του, το καινούριο. Ε, για όλους αυτούς τους λόγους, τους θετικούς λόγους, το σχέδιο έκθεσης που παρουσιάζω έχει μόνο 20 τροπολογίες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν σαν σκοπό να διευκρινίσουν καλύτερα την πρόθεση της ε, πρότασης. Όμως, κάποιες τροπολογίες θέλουν να αναθεωρήσουν το θέμα της εκχώρησης αρμοδιοτήτων προς την Κομισιόν Άρθρο 1 ενώ η Κομισιόν με βάση την πρότασή της προβλέπει μόνο τη χρήση εφαρμοστικών μεθόδων. Εγώ προτείνω να δώσουμε την δυνατότητα στην Κομισιόν να εκδίδει κατεξιδότηση πράξης με βάση τους ορισμούς του περιεχομένου, όχι της δομής του, των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δεδομένων ΑΕ από τα κράτη-μέλη. Καθώς και για τον καθορισμό μέτρων με σκοπό την αξιοπιστία, πληρότητα και συγκρισιμότητα των δεδομένων ΑΕ. Συνολικά, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η Κομισιόν να κάνει μια σωστή διαβούλευση στην προσπασκευαστική φάση και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και αυτές οι διαβουλεύσεις να γίνουν σύμφωνα με την αρχή που υπάρχει στην διαθεσμική συμφωνία του Απριλίου του 2016 για την ε, καλύτερη νόμο Παρασκευή. Για να υπάρχει ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των ε, πράξεων αυτών ζητάω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει παράλληλα με τα κράτη-μέλη και του συμπρόγνωμους των κρατών μελών όλα αυτά τα έγγραφα και να έχει συστηματικά πρόσβαση στι συνεδριάσει των ε, ομάδων εμπειρογνωμών τη Κομισιόν που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατεξιότηση πράξεων. Προσβλέπω στα σχόλιά σα και είμαι έτοιμος να εξετάσω τις τροπολογίες σας. Και τώρα ο κύριος Τόλογιαν από το ΕΛΚΑ, σκιώδης συγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με την αξιολόγησή σας για την χρησιμότητα της πρότασης αυτής της Κομισιόν. Η σημασία του ΑΕ το καθάριστο του εθνικού εισοδήματο δεν είναι μόνο για να υπολογίζει του ιδίου πόρου του προπολογισμού τη Ένωση, αλλά είναι σημαντικό δείκτη για πολλού άλλου λόγου. Για τις διάφορες πολιτικές σε επίπεδο Ένωσης ή σε εθνικό επίπεδο. Φυσικά υπάρχει ανάγκη επικαιροποίηση του κανονισμού με βάση τα επιχειρήματα που μας παρουσιάσατε, Πρόεδρε. Όταν εξετάζω τις τροπολογίες που αναφέρονται και στην έκθεση, μπορώ να πω ότι για τις περισσότερες τροπολογίες ότι είναι πολύ καλές. Εξετάζουμε όμως ακόμα δύο τροπολογίες, δεν έχουμε αποφασίσει. Δημιουργούν κάποια προβλήματα, νομίζω. Μία τροπολογία, η παριθμόν 9, που λαμβάνει υπόψη ότι το GNI, το ΑΕ, υπολογίζεται με τρεις τρόπους. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι υπολογισμού του. Η μέθοδος της παραγωγής, η μέθοδος της χρήσης και η μέθοδος του εισοδήματος. Και στην τροπολογία που προτείνεται, αναφέρετε, εσείς αναφέρετε, ότι μόνο μία μέθοδος θα πρέπει να αναφέρεται στη Eurostat. Νομίζω ότι όμως έτσι περιορίζονται οι πληροφορίες, γιατί κανονικά χρειαζόμαστε και τις τρεις πτυχές για τον καθορισμό του ΑΕ. Και μερικές φορές βλέπεις και τις διαφορές και τις ανακρίβειες που υπάρχουν στο μέγεθος του ΑΕ. Αν, ας πούμε, μία μέθοδος καταλήγει σε ένα ε, ποσό ΑΕ, η μέθοδος, ας πούμε, παρα, παραγωγής ή η μέθοδος, ας πούμε, χρήσης ή μέθοδος του εισοδήματο. Καταλήγει σε άλλα νούμερα για το ΑΕ, κάθε μέθοδος. Και οι τρεις μέθοδοι όμως είναι σημαντικές για τον καθορισμό του ΑΕ. Όχι σε επίπεδο κρατών μελών μόνο, αλλά και σε επίπεδο ένωση. Καλό είναι να έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Φυσικά μπορούμε να το συζητήσουμε. Και είναι και πολύ σημαντική και η άποψη της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Και φυσικά και της Eurostat. Υπάρχει και μια άλλη πρόταση σε αυτή την έκθεση. Απορρίπτει ουσιαστικά μια, την πρόταση της Κομισιόν και είναι η τροπολογία υπαριθμών 14. Η πρόταση της Κομισιόν ε, θέλει να διευκολύνει τη συγκριτική ανάλυση της συμμόρφωσης και γι' αυτό θα πρέπει να κάνει μια απογραφή σε στενή συνεργασία με την ομάδα ε, πυρογνωμόνων που αναφέρεται. Αυτό που κάνουμε με αυτό τον κατάλογο, με αυτή την απογραφή, το κάνουμε για να ξέρουμε σε κάθε κράτος μέλος ποια διαδικασία χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το ΑΕ. Ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω με τον εισηγητή και τους κοιόδες εισηγητές. Για ποιο λόγο εσείς προτείνετε να διαγραφεί αυτή η πρόταση της Κομισιόν. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα και στην αρχή, συμφωνώ πλήρως με τη θέση σας, όπως απεικονίζεται στην έκθεση, καθώς και με την ιδέα για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις ή εφαρμοστικές πράξεις ή εκτελεστικές πράξεις. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση δεν πρέπει να εγείρει πολλά προβλήματα στην Επιτροπή μας νομίζω ότι μπορεί να τύχει πλατιά στήριξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και θα σχολιάσουμε ασφαλώς. Θα σχολιάσω μάλλον ε, η... διαγραφή δεν είναι... το κατάλληλο κατάλογο της υπογραφής. Αμα... Ε, τώρα, από το ECR να ακούσουμε τον κύριο Τσίλερ. Μάλλον, συγγνώμη, μου έστειλε μία ένα σημείωμα ότι δεν μπορεί να παραστεί. Έχει στείλει όμως ένα γραπτό σημείωμα, το οποίο και θα διαβάσω. Τις ευχαριστίες ε, της αφήνω. Το ΑΕ είναι προφανώς ένα σημαντικό μέτρο αμα, μέτρησης και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό τα στατιστικά στοιχεία να είναι τόσο όσο πιο ακριβή γίνεται και συγκρίσιμα μεταξύ κρατών μελών και αυτό περιλαμβάνει και τα πρότυπα και την εναρμόνιση των ημέρων αποστολής. Επίσης τονίζεται η ανάγκη συγκρισιμότητας των δεδομένων παρά τις εθνικές αρμοδιότητες ε, τα ιδιαιτερότητες οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο κύριος Τσίλ επίσης πιστεύει ότι η συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων από τα κρατημέλη εξακολουθεί να είναι κορυφαία σημασία στα πλαίσια της επικουρικότητας, αλλά για να έχουμε και καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα και το, ε, η διαδικασία εναρμόνιση θα πρέπει να συνεχιστεί και υπάρχει ανάγκη να είναι και ενιαία η διαδικασία ελέγχου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προπολογισμού που εξασφαλίζουμε ότι η συνεισφορά των κρατών μελών ελέγχεται και δεν πληρώνει κανείς παραπάνω από το πρέπει ως και ότι του ECR προσβλέπει στη μελλοντική συνεργασία για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ζήλ. Και τώρα δεν βλέπω τον σκιώδη της Άλντα, ούτε της Γκουέ, ούτε και κανέναν άλλον. Άρα να δώσουμε την, ε, το λόγο στον εκπρόσωπο της Eurostat. Ο κύριος Βέμπερ, διευθυντής στη Eurostat και είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Η κυρία μάλλον Βέμπερ, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας προσκαλέσατε σήμερα στην ε, Επιτροπή σα, ό,τι την πρόταση αυτή για τον νέο κανονισμό ΑΕ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον κύριο Κολτιέρη για το σχέδιο έκθεση Η ανάγκη αναθεώρηση του εφιστάμενου νομικού πλασίου προκλήθηκε από τους τρεις βασικούς λόγους τους εξής. Καταρχάς η θέση σε ισχύ του νέου εγχειριδίου ίσα 2010 και το γεγονός ε, ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ορισμοί και οι, τα λογιστικά πρότυπα θα τηρούνται από όλα τα κρατημέλη. Και τρίτον, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κρατημέλη, ότι οι νέες προτάσεις αυτές ε, βοηθούν τη μείωση του φορτίου του παρόχου των ε, στοιχείων στα εθνικα κρατημέλη και στις εθνικές στατικιστικές υπηρεσίες εναρμονίζοντας τις ημερομηνίες για τη χορήγηση των ε, στοιχείων στα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Και είναι σημαντικές οι αλλαγές αυτές, ε, όπως είπε και ο εισηγητής ο κ. Κουαλτιέρη. Σημαντικό είναι άλλωστε και η αλλαγή της βάσης, νομικής βάσης, το άρθρο 338 πλέον, για τους λόγους τους οποίους παρουσίασε ο εισηγητής και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί η παραγωγή των στοιχείων ΑΕ πλέον για σκοπού σκοπούς ίδιων ε, πόρων θα υπάγεται στο πλαίσιο των εθνικών στατιστικών στοιχείων και όλων των σχετικών διατάξεων υπερπιότητας που περιλαμβάνονται σε ό,τι αφορά την, την ουσία. Ο κανονισμός είναι πολύ παρόμοιος με αυτόν που ισχύει σήμερα. Η πρόταση είναι κυρίως τεχνική στη φύση της, με κάποιες διατάξεις οι οποίες ε, ήδη αποτυπώνονται στο σχέδιο έκθεσης της, ε, του εισηγητή που δίνουν ουσιαστικά αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει εναρμόνιση του υφιστάμενου κανονισμού. Προσβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις μελλοντικές συζητήσεις μεταξύ άλλων και των θεμάτων που άπτονται της επιτροπολογίας. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το οικοδόμημα του μοντέλου ίδιων πόρων του ΑΕ όλα τα κράτη-μέλη έχουν φυσικά συμφέρον να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα ΑΕ προκειμένου όλοι να μπορούν να συνδράμουν αυτό που τους αναλογεί στους ίδιους πόρους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είναι σημαντικό να υπάρξουν εφαρμοστικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ακόμα και αν αυτό σημαίνει επιπρόσθετες ε, προσπάθειες από τους παρόχους των δεδομένων. Κλείνοντας, καλώς ορίζουμε την υποστήριξη από πλευράς του Πρόεδρου Γκουαλτιέρη της ευελιξίας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση του κανονισμού και προσβλέπουμε στις συζητήσεις του φακέλου αυτού στις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά τώρα τα παρατήματα. Είναι τεχνική φύσεω και θα πρέπει να καθοριστούν από τους επαγγελματίε στατιστικολόγου. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Είμαστε ασφαλώς στη διάθεσή σας. Εάν επιθυμείτε περαιτέρω διευκρινήσει στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να απαντήσω και σε οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με την αιτιολογική σκέψη υπαριθμών 9. Εγώ έχω να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να το πω και καλύτερα από το είπατε εσείς. Η γύρω στο έχει την εντύπωση ότι χρειάζονται και οι τρεις αυτές προσεγγίσεις για το ΑΕΠ και το ΑΕΠ και αυτό, ξέρετε, δεν αποτελεί καν επιπρόσθετο φορτίο προς τα κράτη-μέλη, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών υπολογίζει και τα τρία αυτά στοιχεία, ακριβώς για τους λόγους που παρουσιάσατε, κυρία Στολογιάν. Πρόκειται για ένα μέσο σύγκρισης και συμφιλίωσης προκειμένου να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή τιμή του ΑΕΠ και του ΑΕΠ. Αυτό λοιπόν τα κρατη το κάνουν ήδη για δικό του συμφέρον και προφανώς θα θέλαμε να λαμβάνουμε και τα τρία αυτά στοιχεία για δικούς μας σκοπούς επαλήθευσης και συγκρισιμότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και συνέβαλαν στη συζήτηση και ασφαλώς με προσοχή θα εξετάσω όλες τις τροπολογίες. να σας ευχαριστήσω για τη σύγκληση που φαίνεται ότι επικρατεί σε ό,τι αφορά την πρόταση. Και εκτιμούμε την ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα μέτρα απογραφής και τα μέτρα σε ό,τι αφορά που αφορούν το περιεχόμενο. Φυσικά θα κοιτάξουμε και τις ε, συμβολέ των συναδέλφων σε ό,τι αφορά τα δύο σημεία που έθεσε ο κύριο Στολογιάννα. Νομίζω ότι επί τη ουσία δεν έχουμε ουσιαστική διαφορά. Είμαι διατεθειμένος λοιπόν να αναζητήσουμε λύσεις για τη διατύπωση. Η τροπολογία νέα τώρα. Σκοπός δεν ήταν να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για ένα και μόνο ζήτημα. Το αρχικό κείμενο δεν είναι και απόλυτα τέλειο. Δεν είναι σαφές τι εννοείται με τις τρεις προσεγγίσεις. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διαφορά επί της ουσίας. Ήθελα απλά να διευκρινίσω περαιτέρω το κείμενο. Αλλά αν πιστεύετε ότι χρειάζεται βελτίωση του κειμένου, να το βελτιώσουμε. Είτε υπάρχει υποχρέωση λοιπόν να παρέχονται και τα τρία στοιχεία, το οποίο δεν το λέει η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή τουλάχιστον ένα από αυτά τα στοιχεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω θα τα βρούμε. Δεν έχω πρόβλημα κανένα να βελτιώσουμε τη διατύπωση. Γιατί 14 θα ελέγξω άλλη μια φορά κατά πόσον ε, δεν λείπει τίποτε. σε ό,τι αφορά δηλαδή τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ πράξεων κατά εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων για τι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσον χρειάζεται κάποια διευκρίνηση. Αλλά ούτε εδώ θεωρώ ότι επί της ουσίας υπάρχει κάποια διαφορά. Σας ευχαριστώ μου λοιπόν και προσβλέπουμε στις τροπολογίε. 22 Νοεμβρίου, η καταλεκτική ημερομηνία, προθεσμία. Μετά θα εξετάσουμε τι τροπολογίε μέχρι τέλη Ιανουαρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Εικόν θα λάβει χώρα φυσικά προς επιβεβαίωση είτε 24 Ιανουαρίου είτε 24 Φεβρουαρίου. Και φυσικά σκοπός μας είναι να πάμε σε τρεμερή διάλογο και να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό το των δυνατών. Δεν φαντάζομαι να μας πάρει πάρα πολύ χρόνο αυτός ο τρομερής διάλογος. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και τους εκπροσώπους της, Ευρωπαϊκής, ε, της και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί η ψηφοφορία προβλέφτεται για τις 17.55. Έχουμε ολοκληρώσει 20 λεπτά νωρίτερα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν και ξεκινάμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στις 17.55 την ψηφοφορία.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 Yeah.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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

Ah.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

Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τις προφορίες μας, ως συνήθως, με μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά, τώρα ηλεκτρονικά. Έναρξη της ψηφοφορίας. όλοι οι συνάδελφοι. Δεν δουλεύει το μηχάνημά σας κύριε Λάγκε. Ίσως τη βάλετε ανάποδα την κάρτα σας. Touch, golden touch. Ε, τι κάνει η γυναίκα, ε. Μαγικά χέρια έχει η γυναίκα πάντα. μαγικά δάχτυλα. Πολύ ωραία. Τελειώνει εδώ η δοκιμαστική ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε με την έκθεση του Φούλβιο Μαρτουσέλο για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης. Συμβασμός A. Υπέρ κατά, άποχες, υιοθετείται. Συμβιβασμός B, υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 52, υπέρ. 53, συγγνώμη διορθώνει ο πρόεδρος, 53. Στο δικό μου κείμενο όμως αναφέρει 52. Γιατί? Πολύ ωραία, να πάρω το σωστό έγγραφο. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε τροπολογία 53 υπέρ. Μου είπαν ότι ο κατάλογος ψηφοφοριών έχει λάθος σειρά. Η γραμματεία μου το λέει αυτό. Οι τροπολογίε 52 και 53 είναι του ίδιου, του κυρίου Βιέγα. Μη σα απασχολεί λοιπόν. Κάνα πρόβλημα. Βασιζόμαστε ε, στο τελικό κείμενο ψηφοφορία. Να πάρω αυτό το κείμενο. Να τσεκάρω και το νούμερο. Ψηφίζουμε τροπολογία 53 υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 53. Ένα ψηφοφορία. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 54 τονικά. Πέρας φοφορίας. Υιοθετείτε. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά. Ελέγχουμε την 55. Πέρας φοφορίας. Υιοθετείτε. Μάλιστα, άρα οι 52, οι 16 και οι 17 καταπίπτουν. Και πάμε στην 17, όχι, στην 56, Πέρα. Στις 56, κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, ένα ψηφοφορία. Ψηφίσουμε τώρα την 56, πέρα ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Με μία ψήφο παραπάνω υπέρ. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τώρα ηλεκτρονικά. Ένα ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Υιοθετείτε. Τροπολογία 58 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 59 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 59, που είναι ένα συνδυασμό. Α, οι σοσιαλιστέ είναι κατά. Μάλιστα, κατάλαβα. Απορρίπτεται λοιπόν, συγγνώμη. Δεν είχα δει καλά τους σοσιαλιστές πώς ψήφισαν. είναι η 59, η 60, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 63 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός C υπέρ κατά αποχές υιοθετείται τροπολογία 78 υπέρ Κατά. Ελέγχουμε την 78. Οι σοσιαλιστές ψηφίσαν. Α, υπέρ. Υπέρ ψηφίσαν οι σοσιαλιστές. Τώρα έχει νόημα να ψηφίσουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Κρατήστε ακόμα την ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άλλοι δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά. Ελέγχουμε την 80. Ένας ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 81 ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 υπέρ, 22 κατά. 82 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 83 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 84 υπέρ. Κατά ελέγχουμε την 84 με ηλεκτρονικό τρόπο. Πέρας Α, ισοπαλία. 21-21. Απορρίπτεται λοιπόν. Πάμε τώρα στην 28. 28. Αιτιολογικές σκέψεις. 28. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την τροπολογία 28. Ηλεκτρονικά. Ενδιαφέρον συνδυασμό των πολιτικών ομάδων. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 29 υπέρ. Κατά. Ας την ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά νομίζω ότι απορρίπτεται. Ψηφίζω τώρα. Πέρας προφορίας απορρίπτεται όντως. 30 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 30. Χρονικά. Περασφοφορία. Υιοθετείται. 32. Το αντίστοιχο τμήμα, corresponding part, 2, υπέρ, κατά, ελέγχουμε 32. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 20 υπέρ, 22 κατά. Συμβασμός D υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 35 υπέρ, κατά. Νομίζω ότι υιοθετείται. Ας την ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε τώρα 35 έναρξη. Πέρας. Υιοθετείται. 36 υπέρ, κατά. Υιοθετείται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά ελέγχουμε την 37. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στην ελέγξουμε εξωτερικά. Έναρξη. Πέρας. Ναι, απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Άποχες δεν βλέπω τους φιλελεύθερους. να ελέγξουμε λοιπόν. Είναι και δική τους τροπολογία στην τελική. Ας τους ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε επί της πρότασης κομισιών, όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα. Ηλεκτρονικά έναρξη. Ακόμα ένα άνθρωπο που δεν ψήφισε. Ψήφισε τώρα. Πολύ ωραία. Κλείνουμε την ψηφοφορία. 39 ψήφι μία ψήφο κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Μαρτουσέλο. Και τώρα πάμε στη δεύτερη. Γραμματεία, πέστε μου ποια είναι. Θα και τον κατάλογο. Είναι η έκθεση της κυρίας Εύα Ζουλή καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων μέσω του ποινικού δικαίου γνωμοδότηση θα του 53 συν τροπολογία υπέρ 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι υιοθετείται ελέγχουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τώρα Vote is closed. Πέρας. Υιοθετείτε. 22 ε, καταπίπτει. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. Υιοθετείτε. 22 υπέρ, 19 κατά. Συμβαστική α υπέρ, κατά, υιοθετείται. Ε, 31 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Συνεχίζουμε. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστικισμός Β, υπέρ κατά ε, αποχές υιοθετήτα. 37, 36 καταπίπτει, 37 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε, 38 καταπίπτει, πάμε στη 39, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40, υπέρ, Κατά αποχές απορρίπτεται 41. Καταπίπτει η 41. 42. Ε, υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 43. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται, 46 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 47 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 48 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 49 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Συμβαστική υπέρ κατά ε, αποχές 53 υπέρ κατά ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. 54 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 55 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 56 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 57 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 58 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 59 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 60 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε, 61 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται, 62 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 63 υπέρ κατά αποχές ε, υιοθετείται, 64 υπέρ κατά αποχές ε, υιοθετείται, συμβαστική ή υπέρ κατά αποχές ε, ε, υιοθετείται, συμβαστική ή υιοθετείται, 64, λήξη, ε, έναξη της ψηφορίας, λήξη. Ισοπολία, άρα απορρίπτεται. 5, υπέρ, κατά έλεγχος. Νομίζω ότι υιοθετείτε αλλά στο ελέγξουμε. Πέρας. υιοθετείτε. 6 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Υιοθετείται. 8 υπέρ. Κατά έλεγχος, έναξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρι... 9 υπέρ, κατά. Έλεγχος, νομίζω ότι απορρίπτεται. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Έναρξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. 11. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έναξη της ψηφοφορίας. λήξη απορρίπτεται. Αυτή ήταν η 12, έτσι δεν είναι. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 10. 15, συγγνώμη. Υπέρ κατά έλεγχος έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική G, υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. Τροπολογία 19. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 20. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφοφορία για την πρόταση της ε, Κομισιόν έτσι πώς έχει τροποποιηθεί. Έναξη της ψηφοφορίας. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένετε. Λήξη. Η 41 υπέρ, 0 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η λήξη η ψηφοφορία, η επόμενη συνεδρία θα γίνει στις, την 5η στις 9, το πρωί, 9 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ.